Mes chers collègues, bonjour. Allez, on va commencer. Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε, λέω, τη συνεδρίασή μα. Έχουμε πολλή δουλειά. Καλημέρα και στου διερμηνεί, λέει η Πρόεδρος. Είμαστε μια χαρά, σα ευχαριστούμε. Ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά. Δεν ξέρω που είναι, λέει, οι Διερμηνεί στη γαλλική ε, ε, καμπίνα διερμηνίας. Χαιρετάει η πρόεδρος. Και εσείς οι Άγγλοι διερμηνείς αισθάνεστε καλά σήμερα. Μπράβο σας. Βλέπω και απέναντί μου τους Φιλανδούς, λέει η πρόεδρος. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Έχουμε Φιλανδούς, έχουμε Σουηδούς. Τέλεια είναι όλα αυτά. Πολύ κόσμο έχουμε. La Hongrie, la Pologne, vous allez bien Et la Roumanie, bien sûr. Ούγγροι, Πολωνοί, Ρουμάνοι, είσαστε καλά. Ξέχασα κανέναν. Η πρόεδρος έχει ξεχάσει τους Έλληνες, αλλά είναι ακριβώ πίσω της η καμπίνα, δεν μας βλέπει. Λοιπόν, όλοι καλά και εγώ καλά είμαι, όπως ακούτε και βλέπετε. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω μια ομάδα εννέα σταζιέρ του, ε, του, της εφημερίδας Μίλτε Μπάιτον Zeitung που έχει καλέσει ο Ισμαέλερ Τουγκ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Εδώ εσείς κρατάτε στα χέρια σας μελλοντική δημοσιογράφοι το μέλλον της, δημο, της ε, δημοκρατίας. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας κύριε Λουκέ. Είστε καλά. L'ordre du jour peut être adopté s'il n'y a pas d'objection. Ε, εγκρίνεται την ημερήσια διάταξη. Πάρα πολύ ωραία. Εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. Πρακτικά των συνεδριάσεων της 19ης και 20ης Φεβρουαρίου 2018 όπως και της συνεδριάσεως της 5 5η Μαρτίου 2018 ε, θα εγκριθούν αν δεν υπάρχουν σχόλια και αντιρρήσεις. Δεν έχω ανακοινώσει από την πλευρά τη Προεδρείου. Μην λυπάστε, μην κλαίτε, δεν πειράζει. Άλλη φορά θα σα έχω τέτοιε ανακοινώσει. Σημείο 4 τροποποίηση του κανονισμού 1018 του 2008 όσον αφορά τους κοινού κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών δραμών στην κοινότητα. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Κλάουντια Ταπαρδέλ θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, μετά θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις ε, εισηγητές και μετά θα ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν και εφόσον έχει εκπρόσωπο, να πάρει το λόγο. Α, καθίσατε αλλού, είσαστε απέναντί μου τώρα εκπρόσωποι της Κομισιόν. Καλύτερα, σας βλέπω πιο καλά. Σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο, κυρία Ταπαρδέλ. Έχετε το λόγο κυρία εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολλοί αυτοί ε, που εργάζονται στην αεροπορία και στα ε, αεροδιαστημικά και θα ήθελα να στείλουμε μία ε, ευχή και μια σκέψη σε αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων που δουλεύουν στον τομέα αυτό γιατί σήμερα είναι η μέρα τους είναι ε, η μέρα που ε, θυμόμαστε και τους κοσμοναύτες, αστροναύτες, καθώς επίσης και τους χιλιάδες ανθρώπους ε, που μας γυρίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, θα ήθελα όσον αφορά το δικό μας θέμα, την τροποποίηση του κανονισμού 10.08 του 2008, να ευχαριστήσω λίγο τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τις οποίες έχουν υποβάλει. Κατανοώ βεβαίως την ε, ε, επιθυμία της Κομισιόν να ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήματα και οι συμφωνίες με τις, με τις Ηνωμένες Αλλά ξέρετε ότι ε, εμείς πρέπει να συζητήσουμε ενδελεχώς τα θέματα. Έχουν προκύψει μια σειρά προβλημάτων στις συναντήσεις με, τη, με, τις, με τα άλλα συμβαλόμενα ε, μέρα. Ε, το weeklies, δηλαδή η μίσθωση με ε, ε, με προσωπικό είναι κάτι που μας προβληματίζει γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και τα δικαιώματα των, ε, του προσωπικού και τα δικαιώματα των επιβατών καλύπτονται. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις αρκετά αποκλίνουσες οι οποίες διαφαίνονται στις, στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Το, η μία προσέγγιση των συναδέλφων είναι να καλυφθούν όλα τα ε, κοινωνικά ε, ζητήματα των εργαζομένων ε, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στα τεχνικά ζητήματα ε, λαμβάνοντα υπόψη τις ήδη υπογραφήσεις ε, διεθνής συμφωνίας. Έπρεπε λοιπόν να τα συζητήσουμε, να δούμε και το θέμα της συμφωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες, γιατί υπήρχε ήδη μια συμφωνία για απελευθέρωση του weight leasing ήδη από το 2017 διαπιστώσαμε ότι πολλοί συναδελφοί συμφωνούσαν με την πρόταση αυτή και επομένως θα δούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να λυθεί το ή τα τεχνικά προβλήματα αυτά. Όμως η αρχική μου θέση ως εισηγήτρια είναι η ίδια ότι, ότι αυτή η τροποποίηση μπορεί να έχει πολύ κακές ε, επιπτώσεις στις ε, αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, κυρίως δε όσον αφορά τα δικαιώματα τα κοινωνικά των εργαζομένων, αλλά και τα δικαιώματα των επιβατών. Επίσης μπορούμε ε, να θεωρήσουμε ότι, θα ότι ναι, ε, αυτή η διαστηριότητα του way leasing είναι εποχική αλλά κινδυνεύει να χάσει αυτόν τον εποχικό ε, χαρακτήρα της και να γίνει πιο μόνιμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και ε, ε, ε, τροποποίησεις. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε μια μέση λύση μεταξύ των... γιατί η μίσθωση με το προσωπικό έχει γίνει πλέον μια πολύ συνήθις λύση στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο ξεχνάμε πολύ συχνά ε, την προστασία των μισθωτών, ε, τις ε, κοινωνικές τις ε, τους, ε, τα κοινωνικά τους δικαιώματα, δηλαδή δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλιση κλπ. Και επίσης τα δικαιώματα των πολιτών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε ε, να ρυθμιστούν καλά οι μελλοντικέ συμφωνίες με τρίτες χώρες χωρίς όμως να κόψουμε και τα φτερά στη δυναμική της αγοράς. Εάν όμως τα δικαιώματα των εργαζομένων και εάν και τα δικαιώματα κοινωνικά και επαγγελματικά επαγγελματικά, εργασιακά ε, τον, ε, του προσωπικού δεν ε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα, τότε πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε καλά. Αναφέρω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετεί χωρίς να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, υπάρχουν άλλωστε και συμφωνίες ε, με άλλες χώρες, εμπορικές συμφωνίες, εταιρικέ σχέσεις ε, και επομένως χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο ε, άρα θα πρέπει να βρεθούν και αυτές οι συμβιβαστικές λύσεις ε, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ε, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού, τα δικαιώματα των πολιτών, των επιβατών και θα καλύπτουν βέβαια και τις ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους με πρώτο τον κύριο Μπάρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ Συγγνώμη κόρες του Μικαήλ Γκάλερ που δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί συνεδρίαζε στη Λιόν το ΕΛΚΑ, συνεδριάζει μάλλον στη Λιόν το ΕΛΚΑ. Ε, στη Γαλλία, κατά εμάς υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που μπορούσαν να είναι αποδεχτές και δει τροπολογίες που έχουν να κάνουν με αεροπορικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί πριν την 1η Ιανουαρίου του 2008 η προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή έδειξε ήδη ότι υπάρχει υποστήριξη στην ρεαλιστική προσέγγιση από την πλειοψηφία των μελών και σε αυτή τη γραμμή θα θέλαμε να εμείνουμε. Σε ό,τι αφορά τις άλλες τροπολογίες και συγκεκριμένα τροπολογίες της εισηγήτριας με τις οποίες εισάγονται νέα στοιχεία στις ιδεολογικές σκέψεις, αυτές οι τροπολογίες χρήζουν περαιτέρω συζήτηση, διότι δεν είμαστε βέβαιοι ότι προσφέρουν προσθέμενη αξία. Παρ' όλα αυτά είμαστε ανοιχτοί ε, στη συζήτηση, ε, στην προσπάθειά μας ε, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να είναι θετικό, από την πλειοψηφία δηλαδή να υποστηριχθεί η έκθεση και την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα το απόγευμα στις Βρυξέλλες, θα έχουμε και τη συνεδρίαση με την εισηγήτρια και τους λοιπούς σκιώδεις. Ευχαριστώ, λοιπόν Κυρία Φώστερ έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κλάουντια, την εισηγήτρια, και να πω ότι πράγματι είναι μια συζήτηση που έχει ε, καταστεί άκρος πολύπλοκη. Ε, υποτίθεται ότι θα είχαμε μια τεχνική τροπολογία και θα τελειώναμε εκεί. Αν όπως το δει κανείς το πράγμα βαθύτερα, θα διαπιστώσει ότι τελικά μάλλον ε, αυτό το τεχνικό ζήτημα έχει περιπλέξει ιδιαίτερα τα πράγματα και ήταν απεριτό Για δεκαετίες ισχύει αυτή η πλήρη μίσθωση, η μίσθωση δηλαδή ασκάφους και προσωπικού. Ε, εγώ θυμάμαι και στην British Airways ότι παίρναμε αεροσκάφη τη Τρανσάβια κάποια εποχή με αυτού του είδους τη μίσθωση γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στο δικό μας στόλο και αυτό κράτησε κάποια χρόνια. Άρα όταν κάποιος καταφεύγει σε αυτή τη μίσθωση υπάρχουν βάσιμοι λόγοι. Σίγουρα υπάρχει το θέμα της ασφάλειας των επιβατών και της ε, λειτουργίας του αεροσκάφους. Βέβαια, δεν ξέρω να υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι αερομεταφορείς που χρησιμοποίησαν αεροσκάφη νεολογημένα σε τρίτη χώρα υποβάθμισαν την ασφάλεια, σε κίνδυνο είτε την ασφάλεια των επιβατών είτε την παρεχόμενη προς τους επιβάτες της υπηρεσία. Τώρα, φυσικά και όλοι θέλουμε να είναι καλοί κοινωνικοί κανόνες ε, και να τους ε, εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη και οι αερομεταφορείς τους. Ε. Αλλά υπάρχουν λόγοι που υπάρχει πλήρης μίσθωση. Δεν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν συνθήκες δουλείας από, για τους εργαζομένους πληρώματος από μία άλλη εταιρεία τρίτης χώρας. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε χώρες ε, της Ένωσης, μεταφέρει χωρών της Ένωσης. Να προσέχουμε λοιπόν αυτά που λέμε. Γιατί φυσικά και θέλουμε να έχουμε ε, κοινούς, ε, καν, κοινωνικούς, καλούς κοινωνικούς κανόνες, αλλά μην είμαστε εμείς ε, αλαζονικοί και να θεωρούμε ότι έχουν τους καλύτερους κανόνες ούτε θα πρέπει να καθορίζει τις λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ε, συμβάσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καταθέσω μάλλον και τροπολογίε και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία. των ασκαφών. για την προσωρινή περίοδο, όσο μικρή και αν είναι, που ισχύει ε, το καθεστώς πλήρους μίσθωσης ε, ουσιαστικά ε, όπως από την Κα, ε, που πήρε η British Airways κάποια αεροσκάφη μπαίνουν στο σύστημα ουσιαστικά της εταιρεία. Ξεκινά δηλαδή ε, λειτουργίες αντίστοιχες με αυτού του βασικού αερομεταφορία. Άρα ο βασικός αερομεταφορέας ε, αναλαμβάνει ε, τις όλες λειτουργίες Άρα θα συμπεριλαμβάνονται στο FTL, στα OPS ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα τρίτα αυτά αεροσκάφη και τα πληρώματά τους. Ε, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πάντα. Δεν μπορούν να φέρουν ένα αεροσκάφος από μια τρίτη χώρα με το καθεστώ πληρωμίσωση, το οποίο όμως του πληρωμάτου και οι κυβερνήτε του θα εργάζονται με, με διαφορετικού όρου και στηρίζω το Μάικλ Γκάλερ. Να είναι απλό. Άρα να μείνουμε στην τεχνική ε, επικαιροποίηση της Κομισιόν, αν δεν σας πειράζει, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δούμε άλλα πράγματα. Πολύ καλή δουλειά της εισηγήτριας, είχαμε και καλές συζητήσεις. Αλλά να τα βάλουμε τα πράγματα ε, στην ευρύτερη προοπτική. Σίγουρα δεν είναι λογικό και κανείς δεν θέλει να συνεχίζεται παόριστον ε, μια μίσθωση τέτοιου είδους. Ε, γίνεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και για βάσιμους λόγους ευχαριστώ την εισηγήτρια αυτά εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπιλμπάου. Έχετε το λόγο κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλες και όλους. Ε, το συναδέλφο θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητρία για τη δουλειά της και γιατί από τη στιγμή που η Κομισιόν κατέθεσε την πρόταση έχει εργαστεί με επιμονή. Ε, δεν νομίζω ότι θα σας ε, εκπλήξει αυτό που λέμε. Το λέμε ως άλντε ήδη από την αρχή. Θεωρούμε πως πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και αυτό το ζήτημα αυτή τη λύση έπρεπε άμεσα να την εγκρίνουμε. Δεν είμαστε υπέρ του πλήρους ανοίγματο και το έχουμε σχολιάσει αυτό και το έχουμε πει και στην εισηγήτρια πάνω από μια φορές. Συμφωνούμε με την αναφορά στις συμφωνίες που γράφονται ε, από την 1η Μαρτίου του 2008. Θα μπορούσαμε αυτό να το δούμε. Θα καταθέσουμε και την τροπολογία μας. Την έχετε, την έχουμε γράψει και άλλοι συνάδελφοι από άλλε ομάδε. Τώρα, θα ε, μπορούσαμε να αρχίσουμε να λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε το δικαίωμα των καταναλωτών, ε, το πλήρωμα, μα όλα αυτά είναι προφανή. Και στην Επιτροπή μας ε, οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό από τις πολιτικές ομάδες δεν κάνουν και τίποτα άλλο στο Κοινοβούλιο που να προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο αυτό και κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Με μια παγκοσμιοποιημένη εστίαση και και στις συμφωνίες της διεθνής που έχουμε υπογράψει. Τώρα όμως μιλάμε για τεχνικό ζήτημα. Το πρόβλημα είναι, το θέμα είναι τέλο πάντων, Μένουμε στο τεχνικό ή ανοίγουμε το θέμα γενικά. Αν θέλουμε γενική αναθεώρηση του κανονισμού, η Κομισιόν λέει ότι θα μπορούσε να μας παρουσιάσει αργότερα μια πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουν μια επανεξέταση του θέματος. Ε. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε επίση και κάποιες από τις τροπολογίες που ανέφερα σε σχέση με τι συμφωνίε που προηγούνται του 1 Μαρτίου 2008 θα συνεδριάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν θεωρούμε όμως ότι πρέπει να υπάρξει ένα γενικό άνοιγμα. Όπως προτείνεται σε κάποιες τροπολογίες πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Αυτός ο κανονικοσμός δίνει την δυνατότητα να μισθωθούν αεροσκάφη νεολογημένα σε τρίτες χώρες για εποχικές αλλάγκες ή γιατί προκύπτουν τεχνικά ζητήματα ή γιατί υπάρχει έλλειψη πληρωμάτων. Η Κομισιόν λοιπόν μας ζητάει ε, να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες διεθνείς συμφωνίες ή διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών. Αυτό ε, βεβαίως ε, σημαίνει ότι θα γίνουν πιο ευέλικτες κάποιες καταστάσεις, αλλά ε, στο μέλλον ε, και ε, μπορεί να προκύψουν προβλήματα και στο πλήρωμα και τα δικαιώματά του και όσον αφορά τους επιβάτες και τα δικαιώματά της. Γι' αυτό λοιπόν δέχομαι την θέση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ότι δεν θα πρέπει να προκύψουν αλλαγές στο εργασιακό και, λοιπά, και καθεστώς και στα δικαιώματα πληρωμάτων και ε, ε, των επιβατών. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να τηρηθούν οι βασικές αρχές και συμφωνούμε γενικώ με την τοποθέτηση και την έκθεση της κυρίας Σταπαρδέλα. Ευχαριστώ πολύ. Κομισιόν, παρακαλώ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρτετς Μπενέχο. Έχετε το λόγο. Um, thank you very Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να χαιρετιστεί την πρόταση του Κοινοβουλίου με σχέδια την κυρία Ταπαρντέλ που προσπαθεί να βρει λύση στο ζήτημα αυτό. Από την αρχή ήμασταν σαφείς ότι ο στόχος της τροποποίησης αυτής είναι να συμμορφωθούμε με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας οι οποίες απορρέουν από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και να ε, φροντίσουμε να μην υπάρχουν διαφορές ε, στην ευρωπαϊκή και στις εθνικές νομοθεσίες. Γι' αυτό λοιπόν οποιαδήποτε πρόταση προς επίλυση του ζητήματος αυτού είναι ευπρόσδεκτη. Νομίζω πω πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ όλους για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Η εισηγήτρια έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις της. Πράγματι, θα συναντηθούμε με τους σχεώδεις εισηγητές για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Μία προς μία. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά αυτά που έχει πει η Επιτροπή, κατανοώ πως υπάρχουν κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αυτό το παρατηρήσαμε περιμέναμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει αυτά τα προβληματικά σημεία και να μην περάσει το πρόβλημα αυτό στο Κοινοβούλιο. Όμως, εδώ πρόκειται για τον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη και γι' αυτό η λύση επήγει. Είναι τεχνικής φύσεως τα προβλήματα. Δυστυχώς ε, μας μεταφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε εμείς τώρα το έργο να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε. Ε, αναφέρθηκαν στην ε, πρότασή μας τα κοινωνικά δικαιώματα, η προστασία του καταναλωτή, τα δικαιώματα των επιβατών στους διάφορους κλάδους μεταφορών. Η πρόταση της Επιτροπής που έχουμε αναφέρεται πολύ συνοπτικά σε όλα αυτά. Υπερβολικά συνοπτικά ώστε να διασφαλίζει την τήρηση αυτών των κατώτατων προτύπων. Υπάρχουν και άλλες εκθέσεις στις οποίες τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των επιβατών κτλ. αναφέρονται επιγραμματικά μόνο. δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, εφόσον λέμε στην Ευρώπη ότι όλα αυτά τα δικαιώματα είναι τόσο σημαντικά, αφήνουμε τα προβλήματα αυτά μόνο σε επιγραμματικές αναφορές και δεν προσπαθούμε να τα λύσουμε. Σίγουρα δεν είναι μόνο προς το συμφέρον ε, των αερομεταφορών να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, είναι προς το συμφέρον όλων και των επιβατών. Πρέπει να δοθεί επιτέλους μία λύση ε, στο θέμα της ε, πλήρης εκμίσθωσης, του wet leasing. Ο ευρωπαϊκός ε, τομέας των αερομεταφορών σίγουρα επιδέχεται βελτίωση, αυτό είναι δίχως αμφιβολία, όμως δεν είναι δικό, δική μας δουλειά να αλλάξουμε τα πράγματα. Και δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στις εσωτερικές υποθέσεις κάθε ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας το δικό μας καθήκον είναι τουλάχιστον να αναφέρουμε τα προβλήματα και τουλάχιστον να αναφέρουμε πως ε, πρέπει να προασπίζουμε τα δικαιώματα των ε, επιβατών, για παράδειγμα, όπως έχουμε ήδη κάνει στο παρελθόν. Χρειάζεται να διατηρήσουμε κάποια συνέπεια, να μην χάσουμε τις ε, κόκκινες γραμμές και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι συμβαστική διάθεση έτσι ώστε να επιληθούν τα προβλήματα. Αλλά να μην ξεχνάμε τη γραμμή που ανέκαθεν ακολουθούσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ταπαρντέλ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Να υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 25 Απριλίου ε, και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα σε, ε, στο επόμενο ε, θέμα ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα. Καλημέρα σας κύριε Ντεπρέ. Le déploiement de Λοιπόν, εναλλακτικά κάψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Όχι γιατί αφορά το μέλλον της βιώσιμης ε, μετακίνησης ε, ή και κινητικότητας στην Ευρώπη, αλλά γιατί καταλαβαίνετε ότι το θέμα έχει ε, και πολλά παρακλάδια περιβαλλοντικά, ε, σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα αλλά επίσης ε, και σχετίζονται και με το μέλλον και την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς επίσης ε, και την ένταξη της πράσινης ενέργειας στην κινητικότητά μας. Θα δώσω λοιπόν αμέσω το λόγο στον κύριο Ισμαέλ Ερτούγκο, ο οποίος είναι εισηγητής. Έχετε το λόγο κύριε Ερτούγκο. Yes, Mrs. thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την κινητικότητα του μέλλοντος. Πρέπει να λάβει χώρα αυτή η μετάβαση προς τις νέες τεχνολογίες. Και πρέπει να πω ότι όσοι ευρωβουλευτέ ήταν εδώ από την προηγούμενη θητεία θα γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια εκπληκτική πρόταση στα πλαίσια τη οδηγία ε, του 2013 και στην πρόταση αυτή υπάρχουν σαφείς στόχοι με συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένα όρια. Ένα από αυτά τα όρια είχε να κάνει με την ύπαρξη 800.000 σταθμών επαναφόρτησης ηλεκτρικών οχημάτων. Και πρέπει να παραδεχτώ εγώ ο ίδιος ότι η Γερμανία, η χώρα μου, άσκησε τεράστια πίεση για να καταστραφεί αυτή η νομοθεσία και τελικά το πέτυχε. Επίσης πρέπει να ασκήσω κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη το είπα αυτό στην ε, τελευταία σύνοδο στο Στραμσβούργο. Να πω ότι αυτή η ανακοίνωση είναι εντάξει, αλλά δεν επαρκεί. Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται το τι πρέπει να γίνει, όμως δεν αποτελεί αυτό νομοθετική πρόταση. Και είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μια νομοθετική πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρηση της πρότασής της. Τώρα μερικά γενικά στοιχεία για την πρόταση. Να πω ότι όταν διάβασα την ανακοίνωση της Επιτροπής συνειδητοποίησα πως υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα νούμερα της Επιτροπής και στα νούμερα τα οποία έχουμε από τη Γερμανία, για παράδειγμα. Τα εθνικά πλαίσια πολιτικής Σύμφωνα με αυτά, μάλλον, μέχρι το τέλος του 2015 η Γερμανία θα έπρεπε να έχει 6.000 ε, σταθμούς επαναφόρτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Όταν επαλήθευσα τις ε, πηγές από το παρατηρητήριο εναλλακτικών καυσίμων, είδα ότι στη Γερμανία θα έπρεπε να υπάρχουν 25.000 σταθμοί επαναφόρτηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά λοιπόν ανάμεσα στα δύο νούμερα. Και διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες διαφορές και γιατί. Έπειτα, το δεύτερο ερώτημα που έχω είναι αν υπάρχει κάποια εναρμονισμένη μεθοδολογία για τις ε, στατιστικές. Και επίσης, πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτά τα σχέδια. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι υπάρχει ανάγκη μέχρι το 2025 να ε, διατεθούν 28 δισεκατομμύρια ευρώ από τα Ταμεία ε, Συνοχής και το, τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Δεν είναι 28 δισεκατομμύρια επιπλέον. Αναρωτιέμαι λοιπόν ε, πώς θα το καταφέρουμε αυτό χωρίς να ε, έχουμε επιπλέον κονδύλια. Εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε υποβάλει μια ξεκάθαρη πρόταση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ταμείο καθαρής κινητικότητας οι υπολογισμοί μα είναι περίπου ίδιοι με, με αυτούς της Επιτροπής. Υπολογίζουμε γύρω στα 24 δισεκατομμύρια ε, ευρώ και νομίζω πως ε, αυτό το ποσό θα είναι αρκετό για να καλύψει αυτούς τους στόχους. Όμως, ε, σε γενικές γραμμές, συνοψίζοντα θα πω ότι η πρόταση αυτή δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται να ε, δοθούν λεπτομέρειες, τα κράτη-μέλη έτσι καθυστερούν και στο κάτω-κάτω έχουμε χάσει και πέντε χρόνια από ε, αυτά που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ερτούγκ Κύριε Ντέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι ο αρχαιώδης εισηγητής, αλλά εκπροσωπώ τον κύριο Σαλίνη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρόν και επομένως θα διαβάσω τη σημείωση που μου έδωσε. Ο κύριος ε, Σελήνη καλωσορίζει την ε, ανακοίνωση της ε, Κομισιόν γιατί θεωρεί ότι θέτει ένα καλό υπόβαθρο όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη και το θέμα των εθνικών προγραμμάτων που υποβάλλονται από, χώρα, από κάθε χώρα μέλος. Η γενική αίσθηση είναι ότι βεβαίως είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την, ε, τους στόχους που είχαν τεθεί στην ε, οδηγία του 2014 4,5 περίπου χιλιάδες σταθμοί επαναφόρτησης μέχρι το 2020 ε, είναι πολύ μακριά από τους ε, στόχους. Ε, υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη σημαντικών επενδύσεων που θα προωθήσουν αυτού του είδους την τοποθέτηση και επίσης να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν ε, κινητοποιηθεί 600, εκατομμύρια έτσι ώστε ε, να καλυφθούν ε, κάποια προγράμματα και οπωσδήποτε θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια και στο επόμενο πολιετές πρόγραμμα. Ε, η Κομισιόν διασυνδέει τις υποδομές αναλλακτικών καυσίμων ε, με τους στόχους ε, για εκπομπές ιδεξιδίου του άνθρακος από τα επιβατικά και άλλα οχήματα. Αυτό είναι καλό γιατί θα πρέπει να προωθηθούν ε, να προωθηθούν εναλλακτικές ε, μορφές ε, κίνησης των επιβατικών αυτοκινήτων, αλλά οι πολίτες συνδέουν το μέλλον αυτών των αυτοκινήτων με τη δυνατότητα επαναφόρτισης τους και τη δυνατότητα πρόσβασης στα καύσιμά τους. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα εναλλακτικά καύσιμα και όχι μονάχα ο, ο, ηλεκτρισμός και η ηλεκτροκίνηση. Ε, βεβαίως ε, συνεχίζει ο, ο σκιώδης ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με, την εισηγητή, με τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος μιλητής δεν είναι εδώ. Κύριε Μάισνερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω... Ευχαριστώ πολύ κύριε Σμάισνερ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έρτουκ. τώρα είναι η εισηγητής. Ε, πριν ήμασταν αντίστροφα, εγώ ήμουν εισηγήτρια, αυτός ήταν σκιώδης. Θέλω να τονίσω και εγώ αυτά που λέει Ισμαήλ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να γίνει αναθεώρηση της νομοθεσίας όταν δεν έχει εφαρμοστεί ε, πλήρως. Δεν ξέρω, το 2000-2022 ε, δεν έχει έρθει ακόμα, είμαστε στο 2018 γιατί η Κομισιόν όμως δεν έχει προτείνει είναι καμία αναθεώρηση και είμαι και απογοητευμένη σε ό,τι αφορά τη μέχρι τώρα εφαρμογή. Θα πρέπει να σας πω ότι ως Κοινοβούλιο είχαμε ζητήσει ε, και αγωνιστεί για μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξίας, ε, ναυσιπλοεία, το LNG να χρησιμοποιείται μέχρι το 2018, αλλά τελικά δεν περιλήφθηκε κάτι τέτοιο, περιλήφθηκε κάτι άλλο. Διότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα των τριμέρων διαλόγων. Αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Και αυτό οφείλεται στο ότι ενώ έχουμε την ανάγκη για τις ε, απαλλαγή, την απαλλαγή από τι εκπομπέ άθρακα στι μεταφόρε, απ' την άλλη έχουμε και το πρόβλημα των χαμηλών τιμών. Και έτσι ξεχάστηκε το θέμα αυτό. Ε, και η ηλεκτροκίνηση δεν ε, ήρθε πιο γρήγορα σε σχέση με τι υποσχέσει ενδεχομένω. Εγώ νομίζω ότι εμεί είχαμε μείνει πολύ σωστά ανοιχτοί για τι αναλλακτικέ τεχνολογίε και σωστά είπαμε όχι μία μόνο τεχνολογία να επικρατήσει. Βλέπουμε όμω σήμερα ότι μπορεί να είναι της μόδας σήμερα στη Γερμανία ηλεκτροκίνηση για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν ε, και άλλα τα καύσιμα, τα βιοκαύσιμα της τρίτης γενιάς ε, κτλ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες εναλλακτικέ ε, και σίγουρα είναι καλό να έχουμε διαφορετικές υποδομές για τις διαφορετικές αυτές μορφές ενέργειας, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστό όρος, ενέργειας για τις μεταφορές. Επίσης, ότι αφορά τη χρηματοδότηση, με το Connecting Europe υπόθηκε. Θα μπορούσε η χρηματοδότηση να εξασφαλιστεί από αυτή τη διευκόλυνση και υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Το πρόβλημα είναι όμως πόσο τελής, πόσο ημιτελής είναι εφαρμογή και αυτό με από ε, γοητεύει ιδιαίτερα και πραγματικά δεν ξέρω ε, που, ε, ποιος, ε, τι έγινε πρώτα η κότα ή το αυγό είναι η γνωστή ιστορία οι καταναλωτές λένε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες τεχνολογίες δεν τις χρησιμοποιούμε κτλ. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να βάλουμε ε, την πάνω ταχύτητα πλέον, να προχωρήσουμε. Θέλουμε να ε, βελτιωθεί και η κατάσταση της, του αέρα της ατμόσφαιρας. Ίσως θα έπρεπε να ασκήσουμε λίγο μεγαλύτερη πίστη σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι βέβαια και να αλλάξουμε αυτά τα οποία γράφει πλέον ε, η νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Ε, δεν είμαι Νομικό εγώ. Νομίζω η προθεσμία που αναφέρεται είναι το 2020-2022, αλλά ε, η Κομισιόν ε, δεν ε, προχωράει. Θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε αυτές τις υποδομές, να προχωρήσουν οι υποδομές για τα εναλλακτικά καύσιμα. Αλλιώς το στόχο μας δεν τον πετύχουμε και περιμένω με ενπομισία την μεταξύ μας συνεργασία και ελπίζω να ασκήσουμε πιέσεις από κοινού. Merci, Σας ευχαριστούμε κύριε Μάισνερ. Και ο Στέλλερ είναι εδώ, δεν σας είχα δει κύριε Τέιλερ. Τέιλορ εννοεί η πρόεδρος. Είμαι εδώ. Yes, thank you. sorry a little... Συγγνώμη, άργησα λίγο, αλλά είμαι εδώ. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης κομισιών για υποδομέ αλλακτικών καυσίμων. Έχω ένα γενικό σχόλιο και κάποια ερωτήσεις αρχικά. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ ότι χρειάζεται περαιτέρω μέτρα για την επιτάχυνση της μετάβασης Ένωση σε, μια, ε, σε ένα τομέα μεταφορών με ή δυνατόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Αλλά πρέπει να τονίσω και κάτι που πρέπει ο κ. Ερτούγκ και άλλοι όμως βουλευτές ότι αυτό το σχέδιο δράση κομισιών δεν είναι φιλόδοξο, ε, είναι άτολμο και δεν μας πάει και πολύ μακριά. Για να τα πω έτσι και με ορολογία μεταφορική. λέγεται ότι υπάρχουν αρκετοί σταθμοί επαναφόρτησης και ότι δεν φταίνουν υποδομές για το ότι δεν αγοράζονται πολλά ηλεκτροκίνητα οχήματα. Πώς η Κομισιόν το βλέπει αυτό έτσι. Πώς συνδέει ε, την χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ε, με τις υποδομές. Και τέλος, τι έγινε με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας βλέπει η Κομισιόν την ανάγκη να υπάρχουν περαιτέρω ε, εξελίξεις σε έναν μόνο τομέα ή και όχι σε περισσότερους ε, τομείς ανακτικών καυσίμων και εάν ναι σε έναν δηλαδή γιατί και σε ποιον κλάδο Κύριε Λουκασέγκα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα. Αυτό ισχύει και για τη δική μου χώρα, η οποία υποφέρει από μεγάλη ε, ατμοσφαιρική ρήπανση και ήδη ακούσαμε πολύ, πολλές φορές ότι υπάρχει θέμα υποδομών. Στην Αυστρία, μια τόσο μικρή χώρα, υπάρχουν ήδη 4.000 σταθμοί επαναφόρτηση, ενώ στην Πολωνία μόνο 600 αυτή τη στιγμή. Και αν μιλάμε για πλήρη σταθμούς που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, μόνο 150. Αλλά να πω πως δεν ε, αρκεί να υπάρχουν μόνο ε, ε, σωστές υποδομές, πρέπει να υπάρχει και η θέληση από τους καταναλωτές να αγοράσουν αυτά τα οχήματα. Και οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ηλεκτροκίνητα οχήματα. Και στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα. Χρειάζεται να ανέβουν οι μισθοί 300% για να μπορέσει ένας καταναλωτής να αγοράσει ένα τέτοιο όχημα. Είναι πάρα πολύ ακριβά αυτά τα οχήματα. Υπάρχουν λοιπόν προϋποθέσεις. Και φυσικά δεν αρκεί μόνο να έχει κάποιο την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα τέτοιο όχημα, πρέπει να μπορεί και να το φορτίσει αρκετά συχνά. Και έτσι λοιπόν μπαίνουν στο παιχνίδι και οι κατασκευαστές αυτών των οχημάτων, οι κατασκευαστές της ε, μπαταρίας. Υπάρχει μεγάλη αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος με τη βιομηχανία, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το μεταβατικό στάδιο, χωρίς να χάσουν τη δουλειά τους ε, άνθρωποι, χωρίς να αλλάξει ριζικά ε, η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και έχω την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορείτε να το καταφέρετε όλο αυτό, ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, πώς ε, θα μπορέσει ένας ε, καταναλωτής να αγοράσει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να μιλάμε για υποδομές. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάννα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ερτούκ και να τον ευχαριστήσω για την τοποθέτηση που έχει πάρει στην ε, έκθεσή του ε, που χρειάζεται βέβαια και κάποια ε, ριζοσπαστικότητα κατά κάποιο τρόπο γιατί και η βιομηχανία και κυρίως μετά από το πρόβλημα που αντιμετώπισαμε με τη Volkswagen και το Diesel είναι σημαντικό να μπούμε πλέον τελειωτικά σε, σε τελική φάση δηλαδή σε κατασκευή αυτοκινήτων με εναλλακτικά καύσιμα και ηλεκτροκίνητα φυσικά είναι αυτονόητο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα της επαναφόρτισης. Γι' αυτό, όπως λέει και ο εισηγητής, χρειάζονται τοποθετήσεις ρίζοσπαστικές όπως αυτές του κυρίου Έρτουγκ. Θα ήθελα ε, να ε, ε, ρωτήσω από την Κομισιόν, ξέροντας βεβαίως, γνωρίζοντας πόσο ανοιχτό πνεύμα έχει και γνωρίζοντας ότι πολλοί εδώ στην Επιτροπή μας είναι πολύ πιο διστακτικοί από την Κομισιόν, εάν απέναντι σε αυτό που είπε και η κυρία Λουκατσέσκα, δηλαδή απέναντι ε, στην, ε, στα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους χρήστες, στους αγοραστές, ε, εάν συζητά για θέματα φορολογικά. Δηλαδή, εάν η Κομισιόν συζητάει και έχει στα ενδεχόμενά της και το θέμα της, των φορολογικών κινήτρων ή ας πούμε το θέμα της μετάβασης από το ένα είδος οχημάτων στο άλλο εάν θα δοθούν κάποια κίνητρα για τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να δώσουν μια πνοή, τα οποία μπορούν να κινητροδοτήσουν επίσης ε, το αστικό πλαίσιο γιατί ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν ε, πολύ διαφορετικά, διαφορετικά μέρη στα αστικά κέντρα γιατί έχουμε από τη μία πλευρά ας πούμε στην Βόρεια Ευρώπη Ευρώπη ε, αυτά, αυτές τις γειτονιές ε, με τα ωραία μικρά σπίτια και από την άλλη μεριά στην Νότια Ευρώπη έχουμε τις γειτονιές με τα πάρα πολύ, τις πάρα πολύ ψηλές πολυκατοικίες, πάρα πολλές οικογένειες κτλ. Επομένως ε, ρωτώ ποιο είδος διαλόγου έχει ξεκινήσει για, να λυθούν τέτοια προβλήματα. Επίσης, ε, όσον αφορά τα δίκτυα, τα ευρωπαϊκά ε, δίκτυα, τα οποία θα συζητηθούν ε, στα τέλη Μαΐου. Θα ήθελα να ρωτήσω στον εκπρόσωπο της τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, η ιδέα της πρότασης ενός τέταρτου πυλώνα όσον αφορά ε, την, ε, ε, ένα τέταρτο πυλώνα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σωστά και με συνέργεια τα κονδύλια και από τους προηγούμενους πυλώνες των μεταφορών, της τηλεπικοινωνίας κλπ. Επίσης τώρα και ακριβώς για να υποστηρίξω τα συμπεράσματα των όσων έγιναν ε, στην Γερμανία, όπως είπε και ο κύριος Ερτούγκ, και τα οποία μπορούν να προβληθούν ε, και στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να βρούμε έναν ε, νέο ένα νέο χάρτη όσον αφορά τους σταθμούς επαναφόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά ε, καύσιμα χωρίς να αλλάξει ε, η ε, ουδετερότητα των καυσίμων. Αναφέρομαι σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα υδρογόνου, φυσικού αερίου κλπ. Αυτές ε, οι υποδομές θα πρέπει να είναι συμβατές, θα πρέπει να έχουν διαλειτουργικότητα, ε, θα πρέπει ε, όταν περνάει τα σύνορα κάποιος να μπορεί παρόλα αυτά να συνεχίζει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του, δηλαδή άμα φύγει από την Πολωνία ή αν φύγει από τη Γερμανία να συνεχίσει στην Πολωνία. Και ξέρουμε ότι και στο θέμα των σορευτών και στο θέμα των ε, γεώσεων ε, υπάρχουν καινου, πολλές καινοτομίες. Άρα ο δρόμος είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βενιτουμπερκ έχει το λόγο. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να χαιρετήσω και τους καλεσμένους σας. Είναι τέσσερα, τέσσερι μαθητές λυκείου που ε, σας ακολουθούν λοιπόν και που προέρχονται και από τις ε, γραμμές ε, της ε, δικιάς σας πολιτικής, του δικού σας πολιτικού κόμματος. Πού είσαστε, μη φοβάστε, σηκώστε το χέρι σας να δούμε πού είστε. Α, αυτοί οι νέοι είναι πολύ ντροπαλοί, λέει η Πρόεδρος. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Κύριε αν έχετε το λόγο. Eh, eh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια αυτά. Ναι, οι νέοι θα έχουν λόγο στο μέλλον. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντική αυτό. Είναι δίχως αμφιβολία. Τώρα, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο δράσης. Ε, χρειαζόμαστε πολύ φιλοδοξία για να το πετύχουμε. Έχω σίγουρα κάποιες ερωτήσεις. Ε, να πω καταρχάς πως είμαι εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το σύνολο της ε, αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι το δικό μας σχέδιο έκθεσης ε, βρίσκεται ήδη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ερτούγκ για, το, για τις δικές του προσπάθειες ε, κύριε Πρόεδρε, το υδρογόνο, η... το φυσικό αέριο, οι άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι η ενέργεια του μέλλοντος. Αυτό είναι δίχως αμφιβολία. Όμως χρειάζεται πολύ φιλόδοξη πολιτική, φιλόδοξα σχέδια και εξαιρετικές υποδομές. Υποδομές για την χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υποδομές που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν αυτά τα οχήματα. Νομίζω πως ε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά μέτρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τους ε, καταναλωτές. Αυτό φυσικά συνεπάγεται και επαρκή πληροφόρηση των καταναλωτών ε, για το πού μπορούν να βρουν σταθμούς επαναφόρτησης, για παράδειγμα. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να έχει μεν την διάθεση να αγοράσει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα ή να το έχει ήδη αγοράσει, αλλά να μην ξέρει πού μπορεί να το φορτίσει. Χρειάζεται επίσης διαφάνεια. Διαφάνεια, για παράδειγμα, στις ε, τιμές ε, των καυσίμων, των αναλλακτικών καυσίμων σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Θεωρώ πως, ε, θα, πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση της Επιτροπής για πράξη κατά εξουσιοδότηση και θα ήθελα να μου εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρόταση. Νομίζω πως θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα. Και πρέπει επίσης να προσέξουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την περιαγωγή, για παράδειγμα. Επίσης, να πω πως έχει ήδη ξεκινήσει ε, η διαβούλευση. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχουν ήδη προκύψει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, φιλοδοξία που πρέπει να δείξουμε, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ε, τι σημαίνει ακριβώς φιλοδοξία, συνεπάγεται αυτό επιδοτήσεις, πώς συνδέεται ε, αυτή η φιλοδοξία που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι υποδομές Αυτές θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο πολιτισμό συνομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη νούμερο 2. Αυτά συνοπτικά ε, τα όσα ήθελα να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται μεν φιλοδοξία, αλλά χρειάζεται και καλή συνεργασία από όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν ε, σε την, ε, αυτή τη φιλοδοξία να πάρει σάρκα και οστά. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Νιτεμπέρκε. Η κυρία Γκονζάλες έχει το λόγο. Κυρία Γκονζάλες παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για την ομάδα μας βεβαίως ε, αυτό το θέμα είναι θεμελιώδους ε, σημασίας. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να, ε, ξεκι... να προωθηθεί αυτό το πρόγραμμα για, τις για τα εναλλακτικά καύσιμα. Να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν είναι ίδια όλα τα εναλλακτικά καύσιμα, δεν έχουν όλα τον ίδιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο ε, αυτά τα καύσιμα τα οποία ονομάζουμε εναλλακτικά. Το ε, το ε, φυσικό αέριο το οποίο το φέρνουμε ε, μετά από χιλιόμετρα αγωγών και που έχει εξαχθεί ε, από μια χώρα που δεν ξέρει τι σημαίνουν κοινωνικά δικαιώματα είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο εναλλακτικό καύσιμα. Κατά την άποψή μας θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να επιλέξουμε εναλλακτικά καύσιμα τα οποία προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας για να είναι πραγματικά εναλλακτικά καύσιμα ε, ε, αν δούμε στις μεγάλες πόλεις ας πούμε, που έχουμε τις περισσότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε αλλαγές στις δομές ε, της ηλεκτροδότησης και μετά θα πρέπει εκτός από το ίδιο το καύσιμο να δούμε και άλλα στοιχεία. Όταν μιλάμε για μεταφορικά μέσα ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν ας πούμε μέσα τα οποία λιγότερο μολύνουν, όπως είναι η, όπως σιδηροδρομικές μεταφορές, άρα θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης ε, την ε, κοινή χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων ή την κοινή χρήση ταξί. Έτσι θα μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν αφορούν ακριβώς την δική μας Επιτροπή και που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρισμού. Αυτός ο ηλεκτρισμός ε, ας πούμε ε, ε, μπορεί να προέρχεται από την καύση στοιχείων στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Εν πάση περιπτώσει έλεγα ότι θα πρέπει να επιλέξουμε εναλλακτικά καύσιμα τα οποία θα προέρχονται και από εναλλακτικέ ανανεώσιμε πηγέ Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Γκοζάκ. Επόμενο ομιλητή, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν, λέει ο κύριο Ρικέ, για ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο μου φαίνεται σημαντικό. Εδώ και αρκετά χρόνια συζητούμε το, το πρόβλημα των δικτύων ε, εναλλακτικών ε, καυσίμων και ε, ηλεκτρικού. Εν τω μεταξύ όμως άλλαξαν τα πράγματα, δηλαδή ξεκινήσαμε στην αρχή με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχαν αυτονομία περίπου 100, 120, άντε 130 χιλιόμετρα. Τώρα φτάνουμε με αυτοκίνητα τα οποία είναι αρκετά προσιτά γενικής παραγωγής φτάνουν σε αυτονομία 400 και πλέον ε, ε, χιλιόμετρων και πολύ σύντομα θα φτάσουμε σε αυτονομία 600 χιλιόμετρων. Επομένως ε, αλλάζει τελείως το πρόβλημα ε, δηλαδή ε, όταν μιλούσαμε για αυτονομία 100-120 χιλιόμετρα θα έπρεπε οπωσδήποτε ε, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα σε αστικό περιβάλλον να υπάρχουν σταθμοί επαναφόρτησης. Εάν όμως η αυτονομία φτάνει στα 500 χιλιόμετρα τότε αλλάζει τελείως η φύση του δικτύου και μάλιστα με διπλό τρόπο. Πρώτον γιατί δεν χρειάζεται ε, ίδιο δίκτυο σε αστικό περιβάλλον. Δεύτερον γιατί ε, θέτει το, το ζήτημα της ε, επαναφόρτισης στο, σπίτι και το είπε προηγουμένως μια ομιλήτρια ότι δεν είναι ίδιο το πρόβλημα στις πολυκατοικίες, το ίδιο το πρόβλημα στα μεμονωμένα, στις μεμονωμένες κατοικίες. Επομένως προκύπτει η διαφοροποίηση όσον αφορά ε, την, ε, ε, τις υποχρεωτικούς σταθμούς επαναφόρτισης στις πολυκατοικίες. Τέλος, εάν υπάρχει ε, επαναφόρτιση ε, στο δρόμο για πιο μεγάλες διαδρομές και κυρίως διασυνοριακές, ε, τότε μπορεί να, να επιλεγεί η γρήγορη επαναφόρτιση. Γιατί αν κάνω ας πούμε μια διαδρομή χιλίων χιλιόμετρων δεν πρέπει να χάσω και τρεις ώρες απλώς για να επαναφορτήσω το αυτοκίνητό μου. Επομένως τροποποιείται ε, το σχέδιο των σταθμών επαναφόρτισης ε, που ε, πλέον έχει ξεπεραστεί από την δυνατότητα των αυτοκινήτων καθώς επίσης και από τις δυνατότητες επαναφόρτισης των σωρευτών. Η Κομισιόν λοιπόν μια και αλλάζει ε, το τοπίο, αλλάζει η Κομισιόν την πολιτική της ε, όσον αφορά τους σταθμούς επαναφόρτησης ε, και τα δίκτυα γιατί σας λέω ότι το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που θα έχει αυτονομία 500-600 χιλιόμετρων θα είναι πραγματικότητα περί τα τέλη του χρόνου σε παραγωγή σειράς κανονικά νομίζω ότι θα πρέπει να διασυνδεθεί η σκέψη που κάνουμε σήμερα ε, με την ε, συζήτηση ε, για τις κατοικίες και τους υποχρεωτικούς σταθμούς επαναφόρτισης στις κατοικίες. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε το θέμα της επαναφόρτισης και των σταθμών επαναφόρτισης γιατί όλη αυτή η συζήτηση ε, ε, θα αλλάξει, θα αλλάξουν οι όροι τους γιατί αλλάζουν οι όροι για την εκδοκίνηση και τους ορευτές. Ε, ευχαριστώ πολύ και εγώ θα πάρω το λόγο τώρα γιατί έχω πολλές ερωτήσεις για την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, συνάδελφοι, όταν μιλάμε για εναλλαγή, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε καλύτερα στο πληθυντικό για εναλλαγές όλοι σε όλες τις ε, χώρες ε, βλέπουν και θαυμάζουν ε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εγώ δεν νομίζω ότι με μία ε, μορφή ενέργειας ε, θα βρούμε λύση για το μέλλον. Θα πρέπει να μιλάμε ε, για το υδρογόνο, για το ηλεκτρικό, για το φυσικό αέριο, ένα μείγμα. Και επανέρχομαι στον, ηλεκτρισμό. Δεν μπορεί να έχουμε διγλωσία δεν, στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν από τη μία μεριά να έχουμε οδικό χάρτη για τις εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όταν λέμε ότι στις μεταφορές θα πρέπει να έχουμε 12% εναλλακτικές ε, μορφές ενέργειας ενώ ε, στο αυτοκίνητο ας πούμε ή στον ηλεκτρισμό να μιλάμε μόνο ε, για παραγωγή από πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορεί να έχουμε δίγλωσία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βασιστούμε στις πραγματικές ανανεώσιμες πηγές. Δεύτερον, πιστεύω ότι το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων πρέπει να διασυνδεθεί με την υποδομή. Και γιατί το λέω αυτό. Το είπε ο κύριος Πρικέα, αναφέρθηκε στους ορευτές, στις μπαταρίες. Πρώτο πρόβλημα. Όσον αφορά ε, τις αστικές ε, περιοχές. Ε, όταν βρίσκεστε στην Ήπεθρο θα βρείτε σταθμούς υπαναφόρτησης. Όχι, θα τα βρείτε μονάχα ε, στην ε, αστική ε, περιοχή. Ή μάλλον το ε, ε, και θα συμβεί και το ανάποδο. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα γιατί δεν μπορούν να τα επαναφορτήσουν στην Ήπεθρο, θα έχουν και μία διπλή τιμωρία γιατί όταν θα έρχονται με το αυτοκίνητό του με τα ε, παραδοσιακά καύσιμα θα του λέμε, α, δεν τα ορυκτά καύσιμα θα του λέμε δεν μπορείτε να μπείτε στι πόλει γιατί απαγορεύεται. Ε, επίσης, κυρία Γκοζάλες, μιλήσατε για τον πλανήτη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους της ΚΟΠ 21 Γιατί στην ουσία βλέπουμε τα κεντρικά στοιχεία του πακέτου της ενέργειας, αλλά δεν βλέπουμε τα παρακλάδια. Σήμερα κανένας δεν μπορεί να αποδείξει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κινείται με ε, ε, ε, πυρηνική ενέργεια μπορεί να ανακυκλωθεί σωστά. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για εναλλαγή εάν δεν μπορούμε να έχουμε και όλο το υπόλοιπο πακέτο της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης. Τέλος, και αυτό αφορά την βιομηχανική πολιτική, δεν είναι δυνατόν να θεσπίσουμε, να θεσμοθετήσουμε τέτοιες τεχνικές εάν δεν θεσπίσουμε ταυτόχρονα και μια νέα βιομηχανική πολιτική. Ποια είναι τα εργαλεία παραγωγή πώ λειτουργούν. Θα σα δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα. Ε, ένα ε, πρατήριο καυσίμων με ορυκτά καύσιμα δεν μπορεί να μεταστραφεί ε, σε, σε σταθμό ηλεκτρικής επαναφόρτησης. Άρα τι κάνουμε με αυτά τα πρατήρια βενζίνης. Δεν μπορούν να ανακυκλωθούν το θέμα μας δεν είναι να βγάλουμε κι άλλα αυτοκίνητα, να παράγουμε κι άλλα αυτοκίνητα. Άρα τι θα κάνουμε με τα αυτοκίνητα τα οποία ε, ε, κυκλοφορούν σήμερα ε, και τα οποία αύριο θα τους πούμε θα πρέπει να μεταστραφείτε και να έχετε εναλλακτικά, να λειτουργείτε με εναλλακτικά καύσιμα. Και επομένως, εάν βγάζουμε αυτοκίνητα τα οποία εξακολουθούμε να βγάζουμε αυτοκίνητα δηλαδή ε, τα οποία είναι παραδοσιακής μορφής ε, και που μολύνουν και μετά λέμε ωραία τώρα θα τα μετατρέψετε τα αυτοκίνητά σας μα αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Εγώ θα μπορούσα να σας μιλάω επί ώρες γι' αυτό αλλά ε, πρέπει να σταματήσω. Κυρία Ντεπρέ έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι να βρίσκομαι εδώ Διότι τελικά τα έχετε καλύψει όλα. Η πρόεδρος διακόπτη. Συγγνώμη κύριε Κράμερ, ήσασταν εγγεγραμμένο στον κατάλογο. Ναι, είχα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Καταρχάς, μιλάμε για εναλλακτικέ ε, τεχνολογίες κίνησης. Αν μιλάμε για τεχνολογία ουδετερότητα τώρα, δεν ξέρουμε τελικά αύριο ε, τι καινοτόμες τεχνολογίες θα έχουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, στη Γερμανία για παράδειγμα, έχουμε μια επιδότηση για το ντίζελ. Τι λέει εδώ η Κομισιόν. Από τη μια πλευρά έχουμε εναλλακτικά καύσιμα και από την άλλη τα παραδοσιακά καύσιμα που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον επιδοτούνται μονίμως. Κάθε λίτρο ντίζελ έχει 18 σέντ του ευρώ επιδότηση, 18 δις ευρώ ετησίως. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά, 8 μάλλον δις το χρόνο, δεν μπορούσαμε να τα επενδύσουμε σε αυτές τις εναλλακτικέ τεχνολογίες και να πούμε όχι. Για επιζή, επιβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον καύσιμα δεν πρέπει να επιδοτούνται, να απαγορευτούν αυτές οι επιδοτήσεις. Έχει να πει κάτι από αυτό η Κομισιόν. Το επόμενο, μιλάμε όλοι για ηλεκτροκίνηση. Το 99% όμως των αυτοκινήτων δεν είναι ακόμα ηλεκτρικά. Για 100 χρόνια έχουμε καταλήξει ε, σε πολύ χαμηλά αποτελέσματα και πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο το ρεύμα. Χρειάζεται πρίζες. Εμείς χαιρόμαστε που έχουμε 13% ενέργεια, ένα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, που ήταν και υπουργό ε, περιβάλλοντος ε, για να σώσει τα εργοστάσια που λειτουργούσαν ε, με άνθρακα ε, έβαλε φρένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς λοιπόν θα στηρίξουμε τα, την αυτοκινητομηχανία σωστά. Αυτό είναι το θέμα και με τα χρήματα των φορολογουμένων. Και για την Κομισιόν ένα ερώτημα. Αν είχαμε 100% ηλεκτρικά οχήματα, όμως στην Ευρώπη να έχουμε 20% μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τι κάνουμε. Είναι καλύτερα τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πρέπει να δούμε τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Και υπάρχουν και έρευνες από επιστήμονες, αλλά δεν ξεκάθαρα. Άλλοι λένε ότι καλύτερα είναι τα βενζινοκίνητα συνολικά σε ό,τι αφορά τον αλυσίδα και τον κύκλο ζωής. Άλλοι λένε είναι χειρότερα. Το θέμα είναι ε, τι κάνουμε αν υποθετικά έχουμε 20% ανανεώσιμες, 80% ε, ενέργεια από κάρβουνο και έχουμε 100% ηλεκτρικά. Εμείς κάνουμε όνειρα τώρα 100% ανανεώσιμες, αλλά κάνουμε σαν να ήταν ήδη πραγματικότητα αυτό. Και μετά από 10 χρόνια μπορεί να έρθει κάποιο ε, και να πει τα σταματώ. Δεν θα έχουμε σε 10 χρόνια 100% ανανεώσιμε. Αυτά τα 8 δι που είπα στη Γερμανία, αν αυτά επιδοτούσαν τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ε, θα βάζαμε αυτή την εισφορά, αυτό το τέλος από 30 στα 50, στα 60, αυτό θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα όμως ε, επιδοτούνται. Ποιος είναι όμως ο συγκεκριμένος στόχος. Ε, ο στόχος είναι να καταπολεμήσουμε τη βλάβη στην υγεία. Σα ευχαριστώ. Τώρα είναι ο λόγος στην κυρία Ντεπρέ. Ευχαριστώ. Τώρα δυσκολεύομαι λίγο πιο πολύ, αλλά τέλο πάντων να ξεκινήσω με το τεχνολο... τα της τεχνολογικής ουδετερότητας. Παρακαλώ, διαβάστε αυτό το σχέδιο, ε, το πρόγραμμα δράση. Είναι τεχνολογικά ουδέτερο. Και θα επανέλθω. Γιατί έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο για τον ε, καταναλωτή. Technological neutral concept εμείς εμένουμε στην αρχή της ουδετερότητας και ιδίως αν δείτε τι κάνουμε με τη διευκόλυνση συνότητα στην Ευρώπη. Συνεχώς προσπαθούμε να επιδοτούμε, να χρηματοδοτούμε προγράμματα που προωθούν τα αναλλακτικά καύσιμα. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την οδηγία σήμερα. Ποιος ήταν ο στόχος της οδηγίας αρχικά. Ήταν να εξασφαλίσει τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών στο δίκτυο τους καταναλωτές. Αλλιώς κάποια κράτη-μέλη θα πίεζαν μία προς μία πλευρά μία τεχνολογία, άλλα σε άλλη κατεύθυνση και δεν θα είχαμε Εμείς λοιπόν δεν έχουμε αλλάξει προσέγγιση. Αυτό θέλω να το πω ξεκάθαρα. Τώρα, πριν πάω στο ίδιο το πρόγραμμα δράσης. να σας δώσω το υπόβαθρο, γιατί δεν έρχεται ε, από τον ουρανό, έτσι ουρανοκατέβατο αυτό το σχέδιο δράσης, γιατί αποφάσισε να καταθέσει δέσμη μέτρων ε, ως πακέτο η Κομισιόν. Είμαστε αυτό, ε, το, σε αυτό το πρόβλημα, κότε το αυγό, εκεί είναι το θέμα. Όμως δεν είναι το μόνο στατικό αυτό. Είπατε αρκετά από εσάς τι κάνει η βιομηχανία με τα οχήματα. Εκεί τι γίνεται. Έχουν καταθέσει μια πρόταση να από το γάμα Δελτα Κλίμα σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα. Όταν εμείς επεξεργαστήκαμε αυτό το σχέδιο πολιτικών και ξεκίνησε και ο διάλογος με τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη λένε ότι τα σχέδια αυτά δεν καταρτίστηκαν ίσως ε, με πάρα, μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση και προσοχή, θα χρειαζόταν ίσως περισσότερο διάλογο. Um, και έρχομαι στον κύριο Ερτούγκ. Τα ίδια θέλουμε κι εμείς. Πιο μεγάλο επίπεδο φιλοδοξίας. Αυτό είναι σαφές. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν τώρα είχε στόχους. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τι έγινε με αυτούς τους στόχους. Είναι τόσο κακά τα πράγματα σήμερα. Σίγουρα δεν έχουμε πετύχει αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, θα έλεγα. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει από την αρχή, καταθέτοντας μια άλλη πρόταση, να την διαπραγματευόμαστε με εσά, με το Συμβούλιο. Πόσο χρόνο θα μας είχε πάρει κάτι τέτοιο, δύο-τρία χρόνια τουλάχιστον. Άρα την ίδια συζήτηση θα μπορούσαμε να την κάνουμε σε τρία χρόνια. Γιατί όταν κάποιος ξεκινά και σχεδιάζει ένα νέο σχέδιο στρατηγικής, στα κράτη-μέλη δεν αλλάζει τίποτα, business as usual. Εμείς λοιπόν είπαμε όχι, ώρα για δράση. Ώρα να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Αναλύσαμε λοιπόν τα σχέδια και νομίζω ότι η προθεσμία που δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία ήταν, πάντως ήταν σίγουρα κάποια είναι τον Νοέμβριο του 2016. 16. Αναλύσαμε τα σχέδια και από τα αναλύσαμε. Ξεκινήσαμε άμεσα διαδικασίες επί παραβάση. Δύο μήνες μετά πήραν επιστολές και θα συνεχίσουν να πέρα επιστολές τα κράτη-μέλη που δεν τα κάνουν σωστά, που δεν εφαρμόζουν σωστά την οδηγία κτλ. Και η διαδικασία συνεχίζεται και την παρακολουθούμε. Αν είμαστε στο σωστό δρόμο για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Θα κάνω μια διάκριση. Τι γίνεται μέχρι το 2020 και τι γίνεται μετά το 2020 και το στόχο του 2030. Αν δείτε το σχέδιό μας, το σχέδιο δράσης, λίγο πολύ είμαστε εντάξει με το 2020 θα δείτε. Λίγο πολύ λέω. Δεν είναι όλα εντάξει δηλαδή, σε όλα τα κράτη-μέλη. Τι κάνουμε όμως, πρώτον. Συνεργαζόμαστε πολύ καλύτερα με τα κράτη-μέλη. Road show. Προσπαθήσαμε να δείξουμε στα κρατη ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι εκθέσεις και οι αναφορές, τα εθνικά πλαίσια κτλ. Θέλουμε ευέλικτα εργαλεία. Θέλω να εξελίσσετε κάθε χρόνο το σχέδιο δράσης και το συνδέω και στο σχόλιο του κυρίου Ρικέ που πολύ καλά μας τα είπε. Τότε είχαμε κάνει μια μελέτη αντικτύπου όταν καταθέσαμε την πρώτη. Τώρα το σενάριο είναι τελείως διαφορετικό. Και για να είμαι ειλικρινής, ίσως είχαμε και κάνει λάθος όλα ως Τα πράγματα όμως ε, στη βιομηχανία εξελίσσονται, εξελίσσονται μπαταρίες, ιδιοχημάτων, πρέπει να τα δούμε. Υπό διαφορετική οπτική γωνία τα πράγματα. Δύο ζητήματα θέλω να φέρω. Σε ό,τι αφορά τι μακρέ αποστάσει, νομίζω είμαστε καλά, αλλά σε ό,τι αφορά τι αστικέ μεταφορέ, όχι και τόσο. Δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο. Και έχουμε και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στι αστικέ περιοχέ, ε, που ελπίζουμε ε, να έχουμε συμφωνία. Όχι μόνο κατοικισμό, αλλά και για τα κτίρια, όπου υπάρχει η δομή, υποδομή καλωδίωση. Έπειτα η σχέση με την Ήπεθρο, με τι αγροτικέ περιοχέ. Και εκεί καλά μα τα είπατε. Πώ θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα, Για κάποια εθνικά ε, σχέδια πολιτικής φτάσαμε σε μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας. και αναγεωγραφική περιοχή. Δεν γίνεται παντού το ίδιο όμως. Πρέπει λοιπόν να γίνουν περισσότερο Χρηματοδότηση, αντιδράσεις και προβληματισμός για το μέλλον. από ο κ. Στέιλορ. την άτολμο το Μην είστε τόσο αυστηρό. Θα σας πω γιατί δεν πρέπει να είστε τόσο αυστηρό. Για πρώτη φορά με αυτό το σχέδιο δράση βλέπετε να συνδυάζουμε πολλές διαφορετικές πηγές και εργαλεία για τον ίδιο στόχο. Το ΣΕΦ, Μα όδησαν και σαν αυτό το γάμα τελτα, 800 εκατομμύρια ευρώ Είχαμε ανακοινώσει κάποια στοιχεία σε σχέση με τις ανάγκες μας για το 2025 και θα πει κανείς ψίχουλα είναι αυτά τα 800 εκατομμύρια. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Και αυτό θέλω να το συνδέσω και με τα σχόλια της κυρίας Αγιάλα. Μίμη, θέλουμε τέταρτο πυλώνα στο πλαίσιο του ΣΕΦ. δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να βάλουμε ε, στη καινοτομία, σε αυτό το σκέλος, ε, περισσότερα κονδύλια τα εναλλακτικά καύση. Χρειάζεται να γίνει αυτό που πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για να αντιμετωπίσουμε και άλλα θέματα που έρχονται να έχουν σημασία με τα εναλλακτικά ή η σχέση με το δίκτυο πάρξης ενέργεια για την ηλεκτροκίνηση. Προκλήσεις σημαντικές, δεν θα πω προβλήματα. Οι νέοι τρόποι για να αντιμετωπίσουν τις μερές προκλήσεις. Οχήματα υποδομές, πώς συνδέονται. Το ευφυές δίκτυο, πώς μπορεί να γίνει πιο ευφυές. Από τη στιγμή που έχουμε περισσότερα στοιχεία από τα οχήματα που περνάνε σε αυτό το ευφυές δίκτυο. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε το χρόνο μας για να σκεφτούμε τι είναι αυτά που χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί στο μέλλον και πώς θα προχωρήσουμε. Σίγουρα όμως με χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Τα στοιχεία. Ότι, δεν υπάρχει, ότι υπάρχει κάποια αναντιστοιχεία. Είπατε κύριε Ερτούκ. Το Φεβρουάριο είχαμε μια επιτροπή που ζήτησε αυτά τα αλλακτικά καύσιμα και το πρώτο που είπαμε ε, στα κράτη-μέλη ήταν ήταν καλά τα νούμερα, σωστά, γιατί δεν παραπονέθηκε κανένα κράτος μέλος. Έχουμε ε, το διάλογο που μας βοηθάει να βελτιώσουμε τα πράγματα. Δεν είμαστε αυθεντοί εμείς. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο σωστά τα δεδομένα. και οι προγραμματικέ δράσει υποστήριξη θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο τη διευκόλυνση τη Ευρώπη σύντομα. Για να γεφυρώσουμε το ΕΤΕΣ για τα ΕΦΗ, ε, τι ΕΦΗ μεταφορέ και για τα αναλυτικά καύσιμα στι δύο κοινότητε, για να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Για να δούμε όχι μόνο τι ε, περιλαμβάνουν τα σχέδια και τα έργα τη Κομισιόν, αλλά και τι γίνεται σε, στην πραγματικότητα. Να δούμε τι γίνεται με τη δημόσια χρηματοδότηση αλλά να δούμε και τι γίνεται με του σταθμού επαναφόρτηση ε, από την ίδια την αγορά. Που χρηματοδοτούνται από την ίδια την αγορά. Και φυσικά και θέλουμε να βελτιωθεί η αγορά ε, ηλεκτροκίνητων οχημάτων από τους να έχουν περισσότερα οχήματα που να αγοράζουν οι καταναλωτές. Τα δεδομένα είναι κάτι σημαντικό αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα οχήματα, ε, αν υπάρχουν σταθμοί, υποδομές, ε, πόσο κοστίζει το ενεργητικό αυτό κάσου κτλ. Μαζί με τα κράτη-μέλη, υπάρχαμε την Επιτροπή Εναλλακτικών, θα, την 3 αύριο και θα μιλήσουν και για τη σύγκριση των τιμών των καυσίμων για να μπορούν οι καταναλωτές να βλέπουν που ε, τους βολεύει και τους ωφελεί τελικά να περάσουν σε ένα εναλλακτικό καύσιμο. Μίλησε κάποιος και για τη διαλειτουργικότητα. Το βλέπουμε. Μπορεί να μην είναι πρόβλημα σήμερα, είναι σημαντικό σημείο και ίσως να γίνει πρόβλημα αύριο. κλείσιμο της αγοράς, ίσως περιορισμό, δηλαδή σε λίγους μόνο οικονομικούς φορείς για τις υπηρεσίες αυτές. Εγώ νομίζω πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε να επαναλάβουμε αυτό που κάνουμε σε άλλους τομείς. Ενεργειακή απόδοση, <clears throat> νομίζω, νομίζω αναφέρθηκα σε αυτή. Ε, κυρία Γιάλα, ε, αυτό που είπατε εσείς είναι αρμοδίδα των κρατών μελών. Όμως, ως μέρος του διαλόγου που θέλουμε να έχουμε με τα κράτη-μέλη. Το θέμα σας το έχουμε ήδη θίξει στο, στα εθνικά πλαίσια πολιτικής και πρέπει να γίνει αυτό, διότι όταν έχεις να κάνεις με την εργαλειοθήκη και με τα κίνητρα, είναι πολύ λογικό, απαραίτητο βασικά, να υπάρχει σωστή σύνδεση των επιμέρους στοιχείων. Ένα λεπτό έχετε ακόμα. Ε, ναι, νομίζω τα κάλυψα όλα. Να αναφερθώ μόνο στο ότι οι προκλήσεις του χθες δεν σημαίνει ότι θα είναι και οι προκλήσεις ε, του σήμερα, του αύριο. Γεωγραφική χρήση του χρηματοδοτικού μέσου, η σύσταση του ίδιου του χρηματοδοτικού μέσου είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, ε, πολύ σημαντική, σημαντικότερη από όλα είναι και η καλή συνεργασία. Κυρία Πρόεδρε, ε, σας καλώ όλους και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής να προσπαθήσετε για όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεπρέ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ώρες, αλλά μας είπατε κάτι σημαντικό. Αυτό που θα ζήσουμε στην αυτοκινητογημανία τα πέντε επόμενα χρόνια δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που ε, ε, ζήσαν οι προηγούμενοι τα προηγούμενα 50 χρόνια και άρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί η επανάσταση δεν θα είναι μονάχα ενεργειακή, ε, θα αφορά και τη συμπεριφορά, θα αφορά τις χρήσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες. Βεβαίως θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, κύριε Ισμαήλ Ερτούγκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ντεπρέ. Νομίζω πως, ε, κυρία Ντεπρέ, υπάρχει επίγουσα ανάγκη να συζητήσουμε. Καλύτερα θα ήταν να το συζητήσουμε και διμερώς, γιατί διαφορετικά ε, νομίζω πως ε, θα ξεχάσουμε πολλά σημεία, θα αποφύγουμε πολλά. τώρα, ε, αυτές οι αναδυστυχίες σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία είναι μια επισήμανση που έκανα και έμεινε απάντητή. Ε, αν έχω καταλάβει καλά αυτά που είπατε, ή έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα με τα εθνικά ε, σχέδια ε, δράσης, ε, τα, η κατάσταση έχει ως Τα κράτη-μέλη δίνουν κάποια στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν αυτά τα νούμερα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, για το υδρογόνο, για το νερό. Υπάρχουν λοιπόν τα στοιχεία που δίνουν, παρέχουν τα κράτη-μέλη και αυτά τα στοιχεία, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση γιατί δεν ε, υπάρχει αντιστοιχεία. Και κάτι άλλο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πως ε, αυτή τη στιγμή ε, δεν αφήνεται τα κράτη-μέλη να τοποθετηθούν, δεν τους αφήνεται περιθώριο. Ε, δεν είχαν τη δυνατότητα να τελέσουν αυτή τη μετάβαση, η οποία μάλιστα προβλεπόταν να γίνει από το 2013. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα όρια και να υπάρχουν και κυρώσεις που θα προβλέπονται όταν αυτά τα όρια δεν θα τηρούνται. Δεν αφήσατε τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, αυτό που έπρεπε, αυτό που ορίζατε. Και τα στοιχεία που έχουμε από τη Γερμανία μας δείχνουν ότι αυτό το πρόβλημα με την κότα και το αυγό θα συνεχίσει να υπάρχει και η κατάσταση κινδυνεύει να επιδεινωθεί. Εμείς ε, ως ε, συνομοθέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το καθήκον να νομοθετήσουμε. Να νομοθετήσουμε πολύ ε, συγκεκριμένα προς το συμφέρον της βιομηχανίας και των πολιτών. Και αυτό αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε και ούτε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όταν υπάρχουν ανακοινώσεις οι οποίες δεν περιέχουν τίποτα το υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη. Και η Κομισιόν εν τέλει είναι και το θεσμικό όργανο το οποίο πρέπει να φροντίσει να ε, πληρούνται οι προποθέσεις, να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Πώς εμείς ε, περιμένετε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις όταν ήδη από την ανακοίνωση με το σχέδιο δράσης μας λέτε ότι μπορείτε να διαθέσετε 8 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μας λέτε όμως καθόλου από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. 800, ε, εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη. Δεν μας λέτε από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αλλά και όχι μόνο, υπάρχει μια τεράστια ε, συζήτηση η οποία έχει περάσει σε επίπεδο συνταγματικών ε, δικαστηρίων και αφορά το πρόβλημα των εκπομπών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο κόσμος έχει αγοράσει αυτοκίνητα με τα οποία εκπέμπουν ρήπους οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα ανώτατα όρια. Και τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημα. Εάν θέλουμε η, βιομηχανία, η βιομηχανία μας να επιβιώσει και πέρα από το 2030 ή το 2040, τότε πρέπει επιτέλους να βοηθήσουμε αυτή τη βιομηχανία να σταθεί και τότε. Αυτό δεν θα γίνει όμως ε, όταν θέτουμε ταυτόχρονα ανώτατα όρια εκπομπών και όταν λέμε ναι θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, θέλουμε να ξεπεράσουμε ε, τα παλιά μοντέλα, να περάσουμε στη, στην ενεργειακή μετάβαση κτλ. Ε, νομίζω πως έχω, έχω μάλλον την αίσθηση ότι δεν ξέρετε τι θέλετε και αυτό ξέρετε περνάει και στην ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Ούτε εκείνοι ξέρουν τι απαιτείται από αυτού. Γι' αυτό λοιπόν εσείς ω ε, συνομοθέτης πρέπει να δημιουργήσετε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο και εμείς θα μπορέσουμε να κινηθούμε. Μόνο εσείς έχετε δικαίωμα πρωτοβουλίας. Και αυτό το άρθρο 10, το οποίο επικαλείστε με το περιθώριο των τριών μηνών, ε, δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει. Εντάξει, μπορεί να σα φαίνονται αρκετά συναισθηματικά φορτισμένα αυτά που λέω, όμως ε, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο εβδομάδων, μηνών, το οποίο ε, υπάρχει, όπου συζητούνται αυτά τα πράγματα και δεν βλέπουμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Εμεί αυτό που θέλουμε επιτέλου είναι μία υποδομή η οποία θα επιτρέψει στη βιομηχανία να ε, φέρει στην αγορά αυτά που απαιτούνται από αυτή. Είτε αυτό αφορά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε. Αυτό είναι το έργο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι δική σας δουλειά να φέρετε αυτές τις προτάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία Ντεπρέ, σας παρακαλώ να συζητήσουμε διμερώς, εσείς και εγώ, για να καταφέρω έτσι να σας μεταφέρω αυτά που προτείνει η δική μου ομάδα και άλλες πολιτικές ομάδες ε, στο Κοινοβούλιο για αυτό το σχέδιο δράσης που παρουσιάσατε. Το ξέραμε ήδη ότι θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Το ξέραμε ήδη από τη στιγμή που το Συμβούλιο αποφάσισε να ε, κάνει κάτι τέτοιο, ότι θα έχουμε τεράστιο θέμα με τις υποδομές. δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τόσο μεγάλες υποδομές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει γονατίσει την ε, βιομηχανία μας. Χάσαμε τρία, τέσσερα χρόνια. Η Κίνα αυτή τη στιγμή ε, κατασκευάζει τρία, τέσσερα εκατομμύρια ε, στήλε επαναφόρτηση θα μπει στην αγορά στο μέλλον, θα είναι η πρώτη δύναμη. Και σε 15-20 χρόνια να είστε σίγουροι ότι τα αυτοκίνητα που θα βρίσκουμε στο εμπόριο θα είναι από την Κίνα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη επειδή δεν δημιουργούμε ένα ε, σαφές πλαίσιο. Δεν θέτουμε ακριβείς στόχους για 20, 30, 40% ε, της, ε, 100. Δεν είναι ε, απαραίτητο να μιλάμε πρώτα για νούμερα χωρίς να υπάρχει πρώτα το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι το σημαντικό γιατί πάνω σε αυτό θα προσανατολιστούμε και θα οδηγηθούμε σε συγκεκριμένες προτάσεις και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν το κάνουμε και δεν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ερτούγκ για αυτό το πάθος με το οποίο μας μιλήσατε και το οποίο ε, είναι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει και την Επιτροπή μας. Σας έλεγα κύριε Ερτούγκ, δεν ακούγατε όμως, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ρόμη με την οποία ακριβώς έχετε αντιμετωπίσει το θέμα, γιατί ε, η Επιτροπή μας με αυτόν τον τρόπο ακριβώς αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν ε, ε, πολύ σημαντικά ζητήματα της δημόσιας υγείας που βρίσκονται στο επίκεντρο όλων. Πάρα πολύ ωραία. Να παραμείνουμε λοιπόν στο περιβάλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας αγαπητοί μου συνάδελφοι και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως διότι υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια ομάδα ε, εργασίας υψηλού επίπεδου που αναφέρεται συχνά σε θέματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για την ομάδα Gear 2030. Gear 2030. Σας καλέσαμε λοιπόν έτσι ώστε να μας πείτε τι συζητάτε μεταξύ σας και να συζητήσετε εδώ, ε, όχι εν κρυπτό και απαραβίστο, αλλά ε, εις το φως της ημέρας και εις επίκον όλων τα όσα θέλετε. Όσοι εγκαταλείπετε την αίθουσα, ησύχως παρακαλώ να την εγκαταλείψετε. Να περιμένουμε λίγο. Si vous sortez, vous sortez πηγαδάκια και συζητήσεις έξω, όχι εδώ. Έλεγα ότι υπάρχει αυτή η περίφημη ομάδα εργασίας ε, και συζητήσεως που θα μας κάνει μια μικρή παρουσίαση ε, και θα ακολουθήσει και ε, συζήτηση. Λοιπόν, όσον αφορά την τελική έκθεση ε, αυτής της ομάδας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δύο χρόνια δημιουργήθηκε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι αυτή η ε, ομάδα εργασίας ε, και εκεί συμμετέχει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας εκπρόσωποι ε, καταναλωτών, ενός ασφάλειας, συνδικάτα και λοιπά καθώς επίσης και ε, πολιτική από την Ευρωπαϊκή και την ε, Εθνική Αρένα, 12 Υπουργοί και 9 Επίτροποι. Αυτή η ομάδα εργασίας ε, είχε στόχο τη διατύπωση στρατηγικών συστάσεων σχετικά με την αντιγωνιστικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά επίσης είχε στόχο τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσεως που αφορά την χρήση και προώθηση των αυτονόμων και αυτοματοποιημένων ε, αυτοκινήτων, εφιών συστημάτων ε, μεταφορών και αυτοκίνητα χωρίς ε, εκπομπές. Το σημαντικό είναι να δούμε θέματα στρατηγικού ενδιαφέροντος για την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η έκθεση αυτή τη ομάδα εργασία ολοκληρώθηκε τα τέλη του 2017 και είμαι ιδιαίτερο ευτυχής που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ για να μα παρουσιάσει συμπεράσματα και συστάσει μετά από αυτήν την ε, παρουσίαση θα έχουμε και την ε, σχετική γνώμη ενός εμπειρογνώμονα του κυρίου Μάσεϊ που βρίσκεστε εδώ Κύριε Μασέ, είστε ε, καθηγητής, ε, καθώς επίσης και αναπληρωτής διευθυντής ε, για, για θέματα κυβερνοασφαλείας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Σας έχουμε καλέσει λοιπόν έτσι ώστε να μας πείτε την άποψή σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δηλαδή. θα δώσω όμως πρώτα απ' όλα τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Κοζίγκου Α, είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα αυτό. Είστε, εκτός του ότι έχετε ωραίο όνομα, είστε και διευθυντής ε, της, ε, ε, του τμήματος ε, βιομηχανικής μεταρρύθμισης και προωθημένων, ασφα, προωθημένων αλυσίδων αξίας από την DigiGrow. Έχετε λοιπόν το λόγο κύριε Κοζίγκου εκπρόσωπε ε, της Κομισιόν. Ε, ναι, είναι ε, το όνομα από τη Βρετάνη και δεν είναι η πρώτη φορά που χαμογελάει κάποιος ακούγοντας ένα βρετάνικο όνομα. Είμαι εδώ λοιπόν για να σας παρουσιάσω ακριβώς αυτά τα θέματα τα οποία είπατε για την ομάδα την οποία αναφέρατε και που είναι γνωστή ως Gear 2030. Όπως είπατε και εσείς, ολοκλήρωσε τον προηγούμενο Οκτώβριο την τελική της έκθεση η ομάδα αυτή. Στόχος της ε, ήταν να προτείνει συστάσεις ε, για την αντιμετώπιση των, κυρίως, ε, των, κυρίων προκλήσεων σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα τον τομέα. Πρόκειται ε, για τους εκπροσώπους αυτοκινητοβιομηχανίας ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό τομέα. 12 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της ε, κινητικότητας 3,3 εκατομμύρια στην αυτοκινητοβιομηχανία και μόνο κατασκευή αυτοκινήτων 90 δις ευρώ εθνικού θετικού ισοζυγίου ε, προκύπτουν από αυτήν την διαδικασία ε, τουλάχιστον μέχρι το 2015 που έχουμε βασίσει τα στοιχεία μας. Ένα σημαντικό τομέα λοιπόν για την οικονομία. Στην τελική έκθεση η εστίαση ανεφέρετο βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, προκλήσεις, ανταγωνιστικότητα, ε, αλυσίδα, αξιακή αλυσίδα, απανθράκωση και τα λοιπά. Απανθρακοποίηση μάλλον και λοιπά. Και ακριβώς εκεί βασιστήκαμε ε, στην ε, μελέτη μας. Ε, θέλω πάντως να αναφέρω κάτι το οποίο είναι σημαντικό γιατί συχνά μας κατηγορούν ότι δουλεύουμε σε σιλό εδώ στην Κομισιόν. Εδώ όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση. Είχαμε επαφές ε, με όλη την ε, αλυσίδα, ε, με τους περιβαλλοντολόγους, με τους καταναλωτές, με την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά είχαμε και την εμπλοκή όλων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέω. Δεν θα πάρουμε τις συστάσεις ε, όλες στη σειρά, ε, γιατί περιμένουμε άλλωστε και μια δέσμη μέτρων από τον επόμενο μήνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 32 είναι οι συστάσεις της Γκίας 2030 ε, γιατί δεν θα προλάβουμε άλλωστε. Έχω όμως ε, να αναφέρω κάποιες από τις προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια καθώς επίσης και κάποια από τα στοιχεία τα οποία θεωρούμε πιο σημαντικά. Επόμενη διαφάνεια. Να πάρουμε πρώτα τις προκλήσεις υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η αξιακή ε, αλυσίδα πιέζεται από πρωτόγνωρες ε, προκλήσεις. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι στα επόμενα πέντε χρόνια θα γίνουν πράγματα που δεν έγιναν τα προηγούμενα 50. Ναι, ε, αναπτύσσονται ε, νέες τεχνολογίες, αυτοματοποιημένη οδήγηση, διασυνδεδεμένη ε, οδήγηση. Αυτό θα σημάνει βεβαίως και πολύ σημαντικές επενδύσεις, αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου, επίσης ε, προσαρμογή σε ε, ε, νέα στοιχεία όπως η αυξανόμενη ας πούμε, χρήση των ε, ρομπότ, μακροχρόνιες βεβαίως, θα, μακροχρό, μάλλον σε μακροχρόνιο ορίζοντα η αυτοματοποίηση θα φέρει οπωσδήποτε θετικά αποτελέσματα, αλλά εντωμεταξύ βράχει πρόθεσμα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Επίσης το θέμα των μηδενικών εκπομπών και της χρήσης αναλυτικών μορφών καυσίμων είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ε, ε, αλλάζουν οι προσδοκίες των ε, ε, των καταναλωτών όλο και περισσότερο μέσω ε, ηλεκτρονικών διαδικασιών αγοράζουν οι καταναλωτές τα αυτοκίνητα, αποφασίζουν να μοιραστούν διαδρομές ε, με άλλους καταναλωτές κλπ. το θέμα της διασυνδεσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία μας αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό ε, και προβλήματα όσον αφορά τα ε, παραδοσιακά αυτοκίνητα. Θα πρέπει βεβαίως να παραμείνει ανταγωνιστική η αυτοκινητοβιομηχανία και άρα χρειάζεται και τη συνδρομή των πολιτικών και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε άλλωστε και η ομάδα υψηλού επίπεδου GEAR το Συμβούλιο ε, λέει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να, υπάρχει, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και ίση δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά. Και αυτό ισχύει και για την βιομηχανία. Επίσης, όλες αυτές οι αλλαγέ θα οδηγήσουν και σε διαρθρωτικές αλλαγέ και σημαντικές αλλαγέ σε ολόκληρες τις φάσεις ε, της ε, ε, αλυσίδα. Υπάρχουν δεξιότητε οι οποίες πλέον είναι παπαλαιωμένες, υπάρχουν άλλε οι οποίες αναδύονται τώρα, Επομένω, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά την κατάρτιση και την επανακατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα η Gear λοιπόν 2030 ε, κάνει κάποιες προτάσεις ε, πρώτα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Είναι σαφές ε, και έχει καταδειχθεί και από το εμπορικό ισοζύγιο ότι ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός τούτη την περίοδο. Η βιομηχανία ε, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή θέση για να παραμείνει ανταγωνιστική. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμα περισσότερο, κυρίως πρέπει να συνεχίσουμε ε, στον τομέα της τεχνικής εναρμόνισης κυρίως στα πλαίσια του φορέα που καθορίζει τα ε, διεθνή ε, πρότυπα. Επίσης να καταπολεμηθεί ε, η τάση προστατευτισμού γιατί και εδώ βλέπουμε και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας βλέπουμε να αλλάζουν οι εμπορικές πρακτικές και να υψώνονται εμπόδια. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες όπως κάναμε μέχρι τώρα και αυτό που θέλουμε στην ουσία είναι να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ένα από τα κέντρα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της παραγωγής αυτοκινήτων. Αξιακή αλυσίδα και δεξιότητες, ο τομέας ε, εξαρτάται ιδιαίτερα από την ποιότητα των προμηθευτών ε, αλλά και ε, από, την, από τις ε, ικανότητες των εργαζομένων. Εμείς έχουμε υποστηρίξει οποτεδήποτε αυτό ήταν απαραίτητο μέσω συγκεκριμένων πολιτικών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, του τομέα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχουν ε, και ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις όσον αφορά ε, το εργατικό ε, δυναμικό και υπάρχουν και κάποια τελευταία γεγονότα τα οποία έχουν αμαυρώσει λίγο τον τομέα. Ε, οι τεχνικές αλλαγές βεβαίως ε, προχωρούν με απίστευτη ταχύτητα και απρόβλεπτη και τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης ε, πολύ συχνά δεν καταφέρνουν να προτείνουν στα παιδιά τις απαραίτητες δεξιότητες. Πολλές λοιπόν τεχνικές συστάσεις έχουν γίνει έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα Erasmus Plus ε, για τα... Είναι το, ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Drives και το οποίο ξεκίνησε ε, το προηγούμενο Ιανουάριο με τετραετή ορίζοντα έτσι ώστε ακριβώς να ε, ε, ε, προωθήσει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στον τομέα της βιομηχανίας, εκπαίδευσης, των σχολείων κλπ. Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθούν οι δεξιότητες που προτείνονται στα κράτη-μέλη, να αναλυθούν αυτές οι προτάσεις σε σχέση με τις ε, μελλοντικές ανάγκες και να καθοριστούν ε, μηχανισμοί συσχετισμού ανάμεσα στην επίσημη και την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση η κατάρτιση είναι απαραίτητο στοιχείο έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στον τομέα. Ε, θα πρέπει επίσης να προβλέψουμε και την αμοιβαία αναγνώριση των καταρτήσεων και αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλη πρόκληση. Ε, θα πρέπει να προωθηθούν άλλωστε και οι διαδικασίες μαθητείας. Υπάρχει και το πρόγραμμα COSME πολύ σύντομα θα δημοσιευθεί και θα έχετε και τις απαραίτητες ε, λεπτομέρειες. Η ιδέα αυτού του project είναι ότι ε, συμπληρώνει ε, το Erasmus Plus δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ταυτοποιήσουν τις επιτυχείς και βέλτιστες πρακτικές. Όσον αφορά τώρα την απαθρακοποίηση και όσον αφορά την εξάρτηση δηλαδή του διοξιδίου του άνθρακα καθώς επίσης ε, ε, και τις μηδενικές ε, εκπομπές υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι μέχρι το 2050 και έχουμε μάλιστα και τη μείωση του 40% μέχρι το 2030. Ο τομέας αυτοκινητοβιομηχανίας βεβαίως τα μάλλον θα συμβάλλει στην επίτευξη αυτή του στόχου και το Gear 2030 ε, κατέδειξε ότι το ρυθμιστικό ε, κανονιστικό πλαίσιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί άμεσα η οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα καθώς επίσης και τα όσα αναφέρονται στο δεύτερο πακέτο κινητικότητας του προηγούμενου Νοεμβρίου της Κομισιόν ε, τα όσα αναφέρονται για τα ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Ε, επίσης, ε, πρόθεση διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων για τις και δημοσίων προμηθειών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η υποστήριξη της μαζικής παραγωγής μπαταριών σωρευτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ορισμένα από τα στοιχεία. Θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα όσον αφορά το σημείο αυτό τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι τεχνολογικός ουδέτερα, αλλά και πρέπει να παραδεχτούμε ότι στον τομέα των μηδενικών εκπομπών τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ε, κατέχουν την ηγετική θέση και αυτό το γνωρίζουν και οι κατασκευαστές. Αναμφισβήτητα, θα, τα επόμενα χρόνια θα ε, αυξηθεί υπερβολικά ε, η ζήτηση των, ε, στον τομέα των μπαταριών. Πολλά στοιχεία λοιπόν πρέπει να προωθήσουμε έχουμε για, τις, ε, για τους ερευτές ε, αυτοματοποίηση, διαδικασίες, ε, δυνατότητα συσσόρευσης κλπ. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι να δούμε τι γίνεται με τα... Asia, China, Korea, Japan. Το σημαντικότερο είναι ότι ε, θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά το θέμα των ε, σοδευτών. Εμείς δεν παράγουμε όλα τα στοιχεία εδώ ε, και είναι σημαντικό να λάβουμε συνολικά υπόψη μας το, το, θέμα γιατί πρέπει να παραμείνουμε ηγέτες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επομένως, ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε είναι να γίνει, να μετατραπεί σε κάτι εμπορικά επιτυχημένο όλη αυτή η καινοτομία και η έρευνα ε, που κάνουμε όσον αφορά ε, τις μπαταρίες. Ε, γιατί μαζί με τις τεχνολογίες που αφορούν τις εκπομπές ε, ε, θα πρέπει να προχωρήσουν πάρα πολύ. Το, τη διετία 19-20 θα δοθεί και ένα εκατομμύριο ευρώ όσον αφορά αυτήν την έρευνα. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της European Battery Alliance που έχει ξεκινήσει τον προηγούμενο Οκτώβριο από τον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Αφού λοιπόν παρουσίασε η γέρα της ε, προτάσεις της. Ε, είναι σημαντικό ε, να υλοποιηθεί η έκκληση του GEAR για υποστήριξη ε, ε, συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων και μεταξύ των projects των εμπλεκομένων όσον αφορά την κατασκευή battery cells. Έχουμε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία γιατί έχουμε ε, ακούσει από πλευράς ευρωπαϊκών εταιριών να αναφέρονται σε δημιουργία ε, ομίλων και για να ακριβώς να προωθήσουν αυτό το ε, θέμα. Η European Battery Alliance ε, είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο καταδεικνύει ακριβώς την ανάγκη προόδου στον τομέα αυτό. Προβλέπουμε ότι θα, προταθούν, ε, και θα προταθεί υποστήριξη και όσον αφορά την κατασκευή και όσον αφορά την ε, ε, εμπορευματοποίηση. Μπορεί να είναι από διάφορους φορείς και διάφορα ταμεία αυτή η οικονομική υποστήριξη. Επίσης, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα μιας βιομηχανικής πρωτοβουλίας, τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά το έχω δει σε τέτοιο εύρος. Είδαμε ολόκληρη την ε, αλυσίδα την αξιακή ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες και να σας πω ότι λαμβάνονται υπόψη και οι πρώτες ύλες καθώς επίσης ε, και τα επίπεδα ασφαλείας ε, της ε, προμήθειας. Και στον τομέα αυτό θα χρειαστούμε νέες δεξιότητες και αυτό αναφέρε, θα αναφέρεται άλλο στο επόμενο, στην επόμενη δέσμη για την κινητικότητα και επομένως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι μπαταρίες θα έχουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά θα είναι και καθαρές γιατί αυτό ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το ανέφερε και η Πρόεδρος προηγουμένω. Όλες οι δράσεις αυτές λοιπόν ε, θα υποστηρίξουν και τις υφιστάμενες εθνικές προτεραιότητες και διαδικασίες στον τομέα αυτό. Ένα άλλο θέμα το οποίο μελετήθηκε από την ομάδα υψηλού επίπεδου GEAR 2030 και είναι το τελευταίο που ανέφερα, είναι τα αυτοματοποιημένα και διασυνδεδεμένα οχήματα υπάρχουν συγκλονιστικές εξελίξεις. Uh, Είπα και προηγουμένως ότι χρειάζεται καλύτερη, ε, καλύτερος συντονισμός των προγραμμάτων έρευνας και των ε, δεξιοτήτων υπογραμμίζεται η ανάγκη δημιουργίας νέων πλαισίων για την υποστήριξη ε, και την υποδομή της των διασυνδεδεμένων αυτών αυτοκινήτων. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη αναθεώρησης των οδικών κωδίκων των χωρών ε, Επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη να αξιολογηθούν ε, σωστά οι μακροχρόνιες επιπτώσεις ε, στις θέσεις εργασίας όσον αφορά δηλαδή τη χρήση αυτών των αυτοματοποιημένων και διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων. Μάλιστα η Ένωση, των, ε, το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών έκανε έκκληση ε, στην ε, Κομισιόν να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θα το κάνει με το, την επόμενη δέσμη κινητικότητα, τον επόμενο μήνα. Θέλουμε στρατηγική η οποία θα διασφαλίζει κεντρικές ε, τεχνολογικές ε, πρόοδους στην Ευρώπη ε, που θα εγγυάται την ασφάλεια των διασυνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων και θα λαμβάνει υπόψη όλη την γνωστή πρόοδο. Επί της βάσεως αυτών των αρχών χρειάζεται βεβαίως και συντονισμένη προσέγγιση και θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα συγκεκριμένοι ε, στόχοι όσον αφορά, και πλαίσιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας, την εμπορευματοποίηση κλπ. και γι' αυτό ακριβώς προκύπτει και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα συνεργατικά και αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα. Κατά την άποψή μας αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ, το θέμα δηλαδή της ύπαρξης ευρωπαϊκής στρατηγικής ε, είναι πολύ ε, σημαντικό και θα συμπεριλαμβάνεται στο, στην τρίτη δέσμη κινητικότητας ε, που θα παρουσιαστεί τον Μάιο. Να σας πω ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η έκθεση της Γκία 2030 ομόφωνα προσυπεγράφει από όλους τους εμπλεκόμενους, πράγμα που δεν το καθόλου πιθανό στην αρχή των συζητήσεων. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους μας. Όπως είπα και προηγουμένως, ξεκινήσαμε ήδη να υλοποιούμε κάποιες από τις συστάσεις και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ε, ίσως θα ήθελε και ο συνάδελφος από την DG Connect να πάρει το λόγο μετά από μένα. Δεν ξέρω αν πώς έχετε προβλέψει. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τη ΓΔ Connect, η δική σας είναι ΓΔ Grow, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Όχι, γάμα δεν move. Έψαχνα. Το ψάχνα, τέλο πάντων. Το βρήκα. Καθηγητά Μάση, για το μέλλον. Καθηγητής ε, και αναπληρωτής διευθυντής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Είστε κατά κάποιο τρόπο προσκεκλημένος εμπειρογνώμονα. Θα έχετε τα λόγο 10 λεπτά για να μας μιλήσετε για τα θέματα αυτά. Καλώ ήρθατε. Thank Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για το θέμα αυτό. Όπως είπατε είμαι στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο αλλά προηγουμένως ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ πάντα για τα θέματα της ασφάλειας υπεύθυνο. Εδώ μιλάμε για τα συνδεδεμένα οχήματα και πώς έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα ασφαλείας και ε, διασύνδεσης υπάρχει πραγματικά μια πραγματική επανάσταση στον τομέα των οχημάτων. Αν δούμε απλά ε, το σύγχρονο software, πάνω-πάνω βλέπετε τους, αριθμ, τους, γραμμοκώδικες σε ένα κανονικό ε, ε, εκατομμύρια γραμμές διπλάσια από την στο facebook στα σύγχρονα αυτοκίνητα και για να μην κάνω σύγκριση με τα διαστημόπλια. Ε, ανέφεραν πολύ ότι λοιπόν ε, εξελίσσεται εδώ η τεχνολογία τώρα για τα αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα. Ήδη υπάρχει αυτή η διασύνδεση, έχουμε αυτές τις ευφύς κοινότητες, αυτά τα δεδομένα δίνουν στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου λοιπά Και υπάρχουν και γεωγραφικά δεδομένα που βρίσκεται, ε, από πού ξεκίνησε και πού πήγε, ε, τι γίνεται με τις θέσεις στάθμευσης, ε, αν πηγαίνει ο οδηγός από το χώρο εργασίας στο σπίτι και αντιστρόφως, περιβαλλοντικά δεδομένα επίσης για τις εκπομπές, την θερμοκρασία, πραγματικά ε, χάρτες ε, ε, με καιρικά με στοιχεία για τον καιρό, θερμοκρασία, από, το, από τους ελοκαθαριστήρες μπορεί να ξέρει κανείς πόσο δυνατή είναι η βροχή, πόσο φυσάει κτλ. κτλ. Ε, είπατε κι εσείς ότι συνδέονται με το FES δίκτυα αυτά τα οχήματα και έχουν επαφή και με πολλά άλλα μέρη. Δεν ξέρουμε και τι άλλες χρήσεις θα υπάρχουν και εγώ που είμαι από την καθημερινή κοινότητα δεν μπορούμε ε, καν να προβλέψουμε εμείς τι γίνεται. Για τα κινητά τηλέφωνα για παράδειγμα κάποιοι λέγανε δεν πρόκειται να πάρουν μερίδιο αγοράς. Φυσικά και δεν έγινε έτσι. Υπήρχαν άλλοι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, μεταξύ άλλων, είχε μιλήσει για την πυρηνική ενέργεια, ότι δεν ποτέ να είναι εφικτή. Πάλι, δεν, ε, πάλι διαψεύστηκε και αυτός. Ε, επομένως δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει το μέλλον, ότι η επανάσταση γίνεται, το ξέρουμε, αλλά πού θα μας οδηγήσει δεν το ξέρουμε. Άρα το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, βοηθήσουμε να υπάρχει περισσότερη καινοτομία. Πώς λοιπόν γίνεται αυτό. Ένα από αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι επειδή δεν ξέρουμε πώ θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα στο μέλλον. Πρέπει να ανοίξουμε την αγορά για την επόμενη γενιά. Φοιτητέ που είναι στο βάθος τη αίθουσα και κάθονται και άλλοι τύποι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τελείως διαφορετικά αυτά τα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να έχουν πρόσβαση στο δεδομένο, να έχουν καινοτόμες ιδέες για να υπάρχει και ανταγωνιστικότητα. Έτσι θα ωφεληθούν και οι ε, παράγοντες ε, που θέλουμε να μπουν ε, στο πεδίο. Θα έχουμε περισσότερη ενέργεια, διαφορετικότητα και φυσικά αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα από τον αυτοκατα... κινητοβιομήχανο και τον κατασκευαστή μέχρι και αυτόν που κάνει καινοτομία να μπορούν να μπουν στο στοίχημα. Έχουμε λοιπόν ανοιχτά πρότυπα επίσης. Όχι για να προβλέψουν τι θα γίνει. Λένε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο αυτοί που καινοτομούν μπορούν να λειτουργήσουν. Για να έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Επίσης θέλουμε κοινά επικοινωνιακά πρωτόκολλα. Έχουμε επικοινωνία μεταξύ οχημάτων. Ε, όλο και περισσότερο στάνταρντ σε ό,τι αφορά την ε, επικοινωνία με την υποδομή, με το χώρο στάθμισης, με τα φανάρια κτλ. Υπάρχει επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Και επίσης ε, υπάρχει επικοινωνία του οχήματος ε, με το σύστημα αυτοματισμού οικίας ή με το κινητό, το FES smartphone που έχουν. Αν μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε με το σύστημα που θα οικοδομήσουμε να προωθηθεί η το θα μας βοηθήσει και στον τομέα της ασφάλειας. Και θα σας μιλήσω για την ασφάλεια των δεδομένων τώρα στο υπόλοιπο που μου, του χρόνου που μου απομένει. Θα έπρεπε να είναι ίσως κάτι δεδομένο για την Κομισιόν, νομίζω είστε και πρωτοπόροι. Μόλις περάσαμε τη φάση που πλέον ε, καταδείχθηκε ότι τα οχήματα είναι ευάλωτα και υπάρχουν ε, απειλές και μάλιστα και επιθέσεις ε, σε αυτά τα οχήματα. Μεγάλη όμως, ε, μεγάλης κλίμακας ε, επίθεση ή κυβερνοεπίθεση οχήματα μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει και ελπίζουμε ποτέ να μην δούμε και να έχουμε μεγάλες τέτοιες καταστροφές. Θέλουμε λοιπόν αποτρεπτικά να δράσουμε. Δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ήδη ε, έχουμε επιδείξεις που μας δείχνουν μπορούμε να κάνουμε στα οχήματα. Στα οχήματα οχήματα ε, αυξάνονται, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία ε, πλέον τα επικοινωνούν τα οχήματα. Και με τον ΚΕΡ 2030 είναι θετικό το ότι αναλαμβάνεται δράση εκ των προτέρων. Εγώ είμαι καθηγητής. Θα σας κουράσω όμως με, μια διαφάνεια που είναι πολύ σημαντική, χωρίς βέβαια να τα ε, πω όλα. Τα και στο Πανεπιστήμιο. Όταν μιλάμε για τις αρχές, πώς θα εξασφαλίσουμε δεδομένα. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το μηδέν, αλλά από αρχές που ήδη ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Θα τονίσω δύο από αυτές. Ε, τον ανοιχτό σχεδιασμό και τη διαχωρισμό του προνομίου. Σε ό,τι αφορά το open design, τον ανοιχτό σχεδιασμό. Είναι σημαντικό στοιχείο ανέκαθεν. Γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί έχουμε να ανταγωνιστούμε έναν ε, εχθρό, έναν αντίπαλο που προσπαθεί να κάνει κάτι κακό στο όχημά μας. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τη δράση του. Εγώ αν είμαι σχεδιαστής του συστήματος δεν είμαι σε θέση να δω με ποιους τρόπους κάποιος θα μπορούσε να επιτεθεί γιατί εγώ το έχω οικοδομήσει αυτό σύστημα και νομίζω έτσι θα λειτουργήσει την άμυνά μου θα τη σχεδιάσω με βάση αυτά που θεωρώ εγώ ότι θα κάνει ο αντίπαλος ε, για να μου τη φέρει. Αλλά οι αντίπαλοι τα σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ και είναι το βασικό πρόβλημα. Είναι μειονέκτημα να θεωρούμε βασικό αναλυτή των κινδύνων τον ίδιο τον σχεδιαστή του συστήματος, γιατί ο αντίπαλος θα σκεφτεί διαφορετικά. Ε, το θέμα είναι ποιες είναι οι προσδοκίες, ε, τι περιμένουμε να συμβεί. Και έχουμε κάνει και πειράματα ε, με εβδομάδε, ε, η μία σχεδίαζε, η άλλη επιτίθετο. Σχεδόν ποτέ δεν συνέβη, σε μένα τουλάχιστον ποτέ δεν συνέβη να έχουν καταλάβει τι θα έκανε η άλλη ομάδα, οι σχεδιαστές. Άρα δεν μπορούμε να το εμπιστευόμαστε αυτό. Θέλουμε λοιπόν ανοιχτό σχεδιασμό και όχι να λέω αναλυτή ο σχεδιαστή θα κάνει αντίπαλο. Πρέπει να έχουν υπόψη ότι κάποιοι μπορούν να σκεφτούν εντελώ διαφορετικά ε, να μα πούνε εγώ έτσι τα επιτιθέμουν. Και όταν όλα αυτά υπόψη. Θέλουμε λοιπόν αυτό το ανοιχτό σύστημα. Τώρα πέραν αυτού του ανοιχτού σχεδιασμού, αυτή η αρχή διαχωρισμού προνομίου, separation of privilege, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ώστε όλα μπορούν να καταλάβουν και να μπορούν να αξιολογήσουν την κατάσταση. Η ασφάλεια μέσω της αδιαφάνειας δεν είναι ασφάλεια Δηλαδή, μόνο αυτό που έχει σχεδιάσει το σύστημα ασφάλεια ξέρει πώ λειτουργεί το σύστημα. Αυτό δεν είναι σωστό τελικά. Τι θα γίνει τελικά. Ο σχεδιαστή και ο αντίπαλο μόνο θα έχουν μάθει πώ λειτουργεί το σύστημα. Καταναλωτέ, διαχειριστή του στόλ, κυβερνητικέ κρατικέ οργανώσει, λόγω διαφάνεια δεν θα καταλαβαίνουν πώ λειτουργεί το όχημα. Όμω οι κακοί θα καταλάβουν πώ λειτουργεί. Θέλουμε λοιπόν πάλι να είναι ανοιχτό ο σχεδιασμό και να υπάρχει πρόσβαση. Δεν θα πρέπει επίσης ποτέ να φανταστούμε ότι υπάρχει περίμετρος ασφαλείας. Κλασικό λάθος να λέμε θα τους κρατάω εκτός οχήματος και δικτύου τους κακούς ή εκτός εταιρεία. Τα έχουμε δει στις ειδήσεις πολλές φορές. Δεν λειτουργεί αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτή η αρχή της, του διαχωρισμού ε, του προνομίου. Δηλαδή κάποια δίστηση μπορεί να υπάρξει στο όχημα, προσπαθώ όμως να τα έχω ξεχωριστά. δεν βάζω όλες τις λειτουργίες ε, στο ίδιο σημείο. Και αυτοί οι διαφορετικοί μηχανισμοί, αυτή η διαφοροποίηση και διαχωρισμός είναι κάτι πολύ θετικό. Αν λοιπόν έχω αυτά τα δύο και δεν λέω ποτέ ότι θα φτιάξω μια, ένα απόλυτα ασφαλέ σύστημα επικοινωνίας για να φτάσει κανείς στο όχημα, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει φτιάξει το τέλειο σύστημα ασφαλείας διότι σφάλουν όσοι μπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν επίπεδα κινδύνων πολύ διαφορετικά και πολύ διαφορετικοί αντίπαλοι που πάντα θα βρουν τον τρόπο τους. Άρα, έχουμε λοιπόν την ανάγκη να έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα με άμυνες. Ίσως μπορεί να, μπορώ να αλλάξω ρεδεφωνικό σταθμό όχημα από κάτι άλλο που είναι πιο δύσκολο. Και κάποιες συστάσεις από την πλευρά σε ασφάλειας. Ανοιχτό σχεδιασμό, Αυτό προωθεί την καινοτομία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αν έχουμε ε, τα σχετικά βέβαια πλαίσια πολιτικής που ενθαρρύνουν ε, τον ανοιχτό σχεδιασμό, την ασφάλεια, την καινοτομία. Όσο πιο ανοιχτό ένα σύστημα, τόσο καλύτερα. Για να μην λέμε ότι εγώ θέλω να προβλέψω τι θα γίνει 5-10 χρόνια μετά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τουλάχιστον εγώ έχω καταλάβει ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη μπορεί να κάνω 5-10 χρόνια μετά θα έχει διαψευστεί και αυτό το βλέπουμε. Και μάλιστα ε, κάποιοι πραγματικά γελιοποιήθηκαν προβλέποντας πράγματα που δεν έγιναν ε, ποτέ έτσι. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργούμε αυτό το σύστημα που θα ευνοήσει και την καινοτομία, το separation of privilege, ε, open design. Είναι σημαντικές αρχές Χαίρομαι για αυτό που κάνετε και επικροτώ τη δουλειά σας για τον ΚΕΡ 2030. Γίνεται τώρα αυτή η δουλειά ε, και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για το ότι μου δώσετε να μιλήσω για όλα αυτά για να προωθήσουμε την ασφάλεια των συνδεδεμένων αυτοματοποιημένων οχημάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μασέ για όλα αυτά που μας είπατε. Ε, ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους έτσι ώστε να ξεκινήσει η πραγματική συζήτηση και θα ξεκινήσω από τον κύριο Ντέλη. Έχετε τον λόγο κύριε Ντέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα, πολλά ακούσαμε και είναι πολλές οι που πρέπει να επεξεργαστούμε. Φυσικά συμφωνώ με το ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ε, στον ηγετικό ρόλο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ελπίζω αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου και το GEAR 2020 να το καταφέρουν αυτό, να κρατήσουν την Ευρώπη στην πρώτη θέση. Τώρα, όσον αφορά την ε, συνδεδεμένη κινητικότητα, που ήταν και το δικό μου σημείο εστίασης, ε, θα ήθελα να πω ότι πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή είναι πολύ επίκαιρο θέμα, είναι επίσης προφανές ότι θα αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Η σχετική οδηγία με κάνει να σκεφτώ την αυτόματη οδήγηση και μετά σκεφτόμουν ότι αν υπάρχει αυτόματη οδήγηση δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την απόσπαση εργαζομένων γιατί τα αυτοκίνητα θα πηγαίνουν μόνα τους. Μέχρι και τα φαρέα οχήματα. Βέβαια, ας φτάσουμε πρώτα μέχρι εκεί και βλέπουμε. Για να φτάσουμε όμως εκεί πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από όλες τις πλευρές. Φυσικά η οδική ασφάλεια είναι ε, μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή όταν γίνεται λόγος για αυτόματα οχήματα. Μετά είναι και το θέμα της, ε, του κυκλοφοριακού προβλήματος, καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιφατικών αυτοκινήτων. Φυσικά όλα αυτά χρειάζονται νέους κανόνες για τους οδηγούς, για την ευθύνη, για τα οχήματα, τις υποδομές κτλ. Χρειάζονται λοιπόν νέοι κανόνες που θα δημιουργηθούν από το μηδέν. Και το θετικό με αυτή την έκθεση είναι ότι προσπαθεί να δώσει κάποιες ε, συστάσεις, κάποιες γενικότερες κατευθύνσεις. Εμείς τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, αλυσίδα αξιών, οφείλουμε όχι μόνο να έχουμε το, στο νου του, την αυτοκίνητο βιομηχανία, αλλά και τους καταναλωτές. Έτσι ώστε όταν ε, ασχολούμαστε με τις νέες τεχνολογίες να μην χάσουμε τους καταναλωτές. Μετά αναφερθήκατε στην τεχνολογία για τις μπαταρίες και είμαι πολύ περίεργος. Τι συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση ε, με τις ε, μπαταρίες ε, solid state. Από όσο γνωρίζω, στην Ιαπωνία έχουν ήδη αρχίσει την ανάπτυξη τέτοιων ε, μπαταριών. Το Ιώτα έχει ήδη μπει δυναμικά στο παιχνίδι. Εσείς λοιπόν πώς βλέπετε τα πράγματα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημάνατε επίσης πως χρειάζονται περισσότερα εργοστάσια, καλύτερες υποδομές ε, κατασκευής μπαταριών. Ε, σίγουρα οι μπαταρίες ε, δεν είναι καθαρή τεχνολογία και αυτές οι καταστάσεις κατασκευής θα εξαρτηθούν επίσης και από το πόσο διαθέσιμες είναι οι πρώτες ύλες, οι οποίες πολύ συχνά προέρχονται από ασταθείς περιοχές. Δηλαδή το κοβάλτι, ας πούμε, προέρχεται από το Κονγκό τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι θα κάνουμε εκεί. Ε, τώρα ε, εξαρτόμαστε από τις ε, χώρες του Περσικού κόλπου για τα ορεικτά καύσιμα. Εξαρτόμαστε από αυτές τις ασταθείς χώρες για ε, τις άλλες πρωτεσίλες. Πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό. Μετά, χαίρομαι πολύ που είχαμε εδώ σήμερα τον κύριο καθηγητή και θα συμφωνήσω μαζί του ο ανοιχτός σχεδιασμός είναι λέξη κλειδί, ιδιαίτερα όσον αφορά τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας. Πώς τα είπατε, δεν θυμάμαι. Ναι, μιλήσατε για διαχωρισμό προνομίων. Τι νομίζετε, σε ποια κατεύθυνση πηγαίνει η αυτοκινητοβιομηχανία. Εγώ πιστεύω πως ε, ίσως πηγαίνει προς αυτό που προτείνετε εσείς, προς τον ανοιχτό συνδυασμό, προς ε, την ε, κυβερνοασφάλεια κτλ. Μη, ή μήπω ε, θεωρείτε πως ε, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες και επειδή όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο σκέψης, τα κλειστά κυκλώματα ασφαλείας λοιπά. Θα υπάρχουν προβλήματα. Εσείς τι γνώμη έχετε λοιπόν γι' αυτό. Πού νομίζετε ε, πώς πηγαίνει η αυτοκινητοβιομηχανία. Ποιος είναι ο τύπος ε, της ασφάλειας που θα χρησιμοποιείτε στο μέλλον. Θα είναι ανοιχτό σύστημα, θα είναι κλειστό. Εσείς τι άποψη έχετε. Αυτά λοιπόν είχα να ρωτήσω. Σας ευχαριστώ. Εξαιρετική ερώτησή σας. Ναι, πρώτα θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και μετά ε, θα έχετε τον χρόνο να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής ε, Πράγματι, η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Περάσαμε το σκάνδαλο με τις εκπομπές ρήπων που αμαύρωσε τη φήμη της, θέματα με την υγεία, με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλάζουν οι προσδοκίες του κοινού και αλλάζει και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Το 2030 είναι μια καλή αφορμή για να ξεκινήσουμε ξανά, να γίνει επανεκκίνηση. Γι' αυτό λοιπόν ε, βλέπουμε πως υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και από τις ε, κυβερνήσεις ε, στην επένδυση σε ηλεκτρικά οχήματα, σε αυτόματα οχήματα. Όμως χρειάζεται και αποτελεσματική υποδομή, αρκετά ευρέως διαδεδομένη. Χρειάζεται επίσης και συνδεσιμότητα, χρειάζεται δίκτυο 4G. Όλα αυτά συνδέονται και με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως με το δίκτυο 5G. Για να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα δικτυωμένα οχήματα που ακούσαμε. Βέβαια, έχουμε φτάσει αρκετά μπροστά. Ε, τώρα τα ηλεκτρικά οχήματα θα διδαματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση της ε, ατμοσφαιρικής ερήπανσης από τον τομέα των μεταφορών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ε, των κατοίκων των πόλεων. Και ως ε, σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα να προσπαθήσει να ε, καταρτήσει αποτελεσματικά σχέδια που θα, έχουν, ε, θα δώσουν έμφαση στην ασφάλεια και την υγεία. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον κύριο καθηγητή εάν συμφωνεί με αυτήν την στενή σχέση ανάμεσα ε, στις νέες τεχνολογίες και στο δίκτυο 5G και, είναι, ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπούτο. Κύριε Κράμερ, θέλετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Πολλές ερωτήσεις έχω, αλλά θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ στα ουσιώδη. Καταρχάς, ποια είναι η εμπειρία σας με το Cars 21 και το Gear 2030. Μπορείτε να μας πείτε πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό την αυτοκινητοβιομηχανία έτσι ώστε αυτή να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος έπειτα. Ε, το ανέφερα και πριν. Ήδη στη Γερμανία είχαμε τις επιδοτήσεις για τα ντίζελ. Ε, αυτά τα αυτοκίνητα είναι πιο... Ε, θεωρούταν ότι καταναλώνουν λιγότερο ντίζελ, λιγότερη ενέργεια και είναι πιο καθαρά. Όμως... Το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Ο συλλογισμό είναι αρνητικό. Με τα ντίζελ καταφέραμε το αντίθετο από αυτό που θέλαμε, διότι βλέπουμε πω σήμερα οι εκπομπέ ρήπων από τα αυτοκίνητα ντίζελ είναι πολύ ψηλότερε σε σχέση με παλιά. Τώρα οι πρωτοβουλίε νομίζω πω πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Για του νέου τώρα δεν είναι πλέον τόσο σημαντικό να βγάλουν δίπλωμα οδήγηση. Όταν ήμουν εγώ νέος ήθελες ένα χρόνο μέχρι να βγάλεις δίπλωμα. Από τα 17 στα 18 και ήθελες διακαώ να βγάλεις δίπλωμα για να πάρεις αυτοκίνητο. Βλέπουμε ότι οι νέοι σήμερα δεν πολυκαίγονται να οδηγήσουν. Δεν τους πειράζει κιόλα. Και αυτό έχει οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των οχημάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις πόλεις βέβαια και θα είναι πολύ ωφέλιμο. Όμως τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι, Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί στηρίζονται ε, στις, ε, στα οχήματα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα τρένα, υπάρχουν και τα πλοία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι μεταφοράς και υπάρχουν άπειροι τομείς που συνδέονται με αυτά. Η παραγωγή ενέργειας, ε, ηλεκτρισμός κτλ. Όλοι αυτοί κινδυνεύουν με χρεοκοπία αν αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα. Εμείς, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο η δική μας επιτροπή ε, αρμόδια δεν είναι μόνο η ε, Επιτροπή Μεταφορών και η Επιτροπή Ήτρε και η Επιτροπή Ίντα η Γραμματεία, διάφορες επιτροπές. Ε, αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα σε πολλά επίπεδα και εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε τα προβλήματα με το κοβάλτιο, ξέρουμε τα προβλήματα με την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, όμως δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τον καταναλωτή, πρέπει να διευρύνουμε την οπτική μας, το οπτικό μας πεδίο και να δούμε το, τη γενική εικόνα. Τώρα, κύριο, υπάρχει ένας καθηγητής, ε, ο καθηγητής Σου στο Άχεν, ο οποίος ε, δημιούργησε, κατασκεύασε μάλλον ένα μικρό φορτηγό ηλεκτροκίνητο. Και ξέρετε τι έγινε. Κανένας δεν ήθελε να το κατασκευάσει μαζικά. Γιατί το κόστος ήταν υπερβολικά υψηλό. Αυτή η τεχνολογία δηλαδή υπάρχει, υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά κανείς ε, δεν θέλει να την εφαρμόσει. Σε αυτές τις ε, επιτροπές λοιπόν αυτό που θα έπρεπε ίσως να συζητηθεί είναι γιατί δεν προχωράμε, γιατί δεν εφαρμόζουμε την τεχνολογία που ήδη διαθέτουμε έτσι ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς ε, τους ε, στόχους που έχουμε θέσει. Τέλος, ε, όσον, αφορά όσον αφορά το σκάνδαλο με τον ντίζελ, εσείς τα ξέρατε, γιατί τι κάνατε τόσο καιρό, γιατί σιωπούσατε. Και μα είπατε ότι δεν γινόταν, δεν μπορούσαμε. Ωραία, ναι. Αν δεν μπορούσατε λοιπόν με όλε αυτέ τι επιτροπέ να κάνετε τίποτα, γιατί τι έχετε τι επιτροπέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Κυρία Κλούν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και τους ε, άλλους ομιλητές ε, για το GR 2003, την έκθεση αυτή. Είναι σημαντικό να δούμε συνολικά στη βιομηχανία πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ίσως παραλαμβάνω αυτά που υπόθηκαν πριν, αλλά μειωμένη χρήση οχημάτων. Το είπαμε. Αν ζουν λιγότερες πόλεις, ε, θέλουμε, ε, θα υπάρχουν και λιγότερα οχήματα. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πάρα πολύ ε, στη, στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς το αντίθετο θα πετύχουμε στις πόλεις, δηλαδή να μην παίρνουν αυτοκίνητα οι άνθρωποι, αλλά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ε, και νομίζω ότι αυτό επικρέματος δαμόκλειο πάθ πάνω από τις αυτοκίνητες μηχανίες και σε ό,τι αφορά την χρήση ε, του ίδιου χήματος από περισσότερους, στο καρσέν κτλ. κτλ. ή κάποια μίσθωση ή κάποια ε, το go-car για παράδειγμα, κάποια τέτοια συστήματα ή η χρηση ποδηλάτων. Και επίσης το πρόβλημα των πρώτων υλών για τους ορευτές, για παράδειγμα χρειάζεται πιο πολύ χαλκός για παράδειγμα για τα ηλεκτρικά οχήματα, αυτό είναι ένα θέμα. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Όσο προχωρούμε θα εξαρτηθούμε από τους σπόρους αυτούς, αλλά δεν ελέγχουμε ε, τα αποθέματα. Πρέπει να το έχουμε υπόψη και αυτό. Να ευχαριστήσω και τον ε, καθηγητή Μάση. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ελπίζω να έχουμε τις διαφάνειες. Ήταν αφήσω όμως και η προσέγγιση που μας παρουσιάσετε. Σε ό,τι αφορά το, το separation of privilege. Η ορολογία σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Μας δίνει ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε τα πιο σημαντικά από τα λιγότερο σημαντικά. Κανείς δεν θα ήθελε να σκεφτεί καν ότι μπορεί κάποιος ε, ε, από απόσταση να πάρει τον έλεγχο του οχήματος και να το χρησιμοποιήσω ως για παράδειγμα. Merci Ευχαριστώ για την κυρία Κλούν και εγώ ως πρόεδρος έχω τις ερωτήσεις μου. Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω τι θα πει ε, αυτό το Gear 2030. Μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου λέτε που εργάζεται πολύ με όλους. Ε, ναι, ωραία. Τι στόχο έχει. Πού υπάγεστε στο Συμβούλιο, ε, έχετε απλά ε, την ε, ε με το να δίνετε κάποιες γνωμοδοτήσεις στην Κομισιόν. τι είστε ακριβώς, ποια είναι η αποστολή σας, είναι ουσιαστικό το ερώτημα. Εγώ την ύπαρξή σας τη γνώριζα, δεν έχω καταλάβει όμως. Εμείς είμαστε νομοθέτες. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνετε εσείς. Εγώ έχω ένα πρόβλημα και δουλειά μου εμένα είναι να μάθω εσείς ακριβώς τι κάνετε. Τι κάνετε μέσα αυτές τις, ε, στα θεσμικά όργανα. Ανήκετε στο Συμβούλιο, ε, στη, στο Κομισιόν, μα λαμβάνονται αποφάσεις. Ε. Επηρεάζετε εσείς πώς, τι γίνεται. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο. Κάποιοι από τους συνάδελφους είπαν και το πανέλαβαν άλλοι ότι θα μειωθεί ο στόλος των οχημάτων στο μέλλον. Έτσι θα γίνει. Τις οικονομικές επιπτώσεις τις έχετε μελετήσει. Άμεσες και έμεσες επιπτώσεις για την απασχόληση. Γιατί το είπατε εσείς, ένα από τα πρώτα στοιχεία είναι 12 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία. Με την ψηφιακή επανάσταση του αύριο θα χαθούν δεξιότητες και θα χαθούν και θέσεις εργασίας, επαγγέλματα. Οι άνθρωποι αυτοί που θα χάσουν τη δουλειά τους και που δεν καταλαβαίνουν τίποτα με, ότι έχει να κάνει με αλγόριθμους, ε, με τα σύμφωνα και τα αυτούς τους ανθρώπους θα τους κάνουμε. Τρίτον, ο κύριος Μάση Μας παρουσιάσετε με αρκετά ευληπτό τρόπο ε, τη σημασία της πρόσβασης στα δεδομένα. Είναι σαν το αυριανό καύσιμο, αν θέλετε, η πρόσβαση στα δεδομένα. Και επιμείνατε στο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στα θέματα της κυβερνοασφάλειας από τους ε, κατασκευαστές. Η ομάδα εργασίας τι κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. δεν θα υπάρχει μεγάλη απειλή για τον ανταγωνισμό. Βλέπουμε start-up εταιρείε που θέλουν να προχωρήσουν και τους λέμε ότι θα κρατάει αυτοκινητοβιομηχανία τα δεδομένα. Αυτή λοιπόν η αφής επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει για άλλες μορφές κινητικότητας. Πώς λοιπόν θα φροντίσουμε να έχουν αύριο πρόσβαση στα δεδομένα και οι νοφείς επιχειρήσεις και τι θα κάνουμε ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα για όλους και όλες να μην οδηγήσει στο εξή. Κάποιοι να κρατάνε τα δεδομένα και έτσι να ε, παρακολουθεί η δυνατότητα καινοτομία. Αυτά εσεί τα έχετε μελετήσει σε εσά κύριε Μάση. Τέταρτη ερώτηση για τον κύριο Μάση πάλι. καλά πάνε τα πράγματα με την ανάπτυξη των ε, αυτόματων οχημάτων, δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις ε, και στο ίντερνετ όλοι πάνω στο αυτόματο όχημα δουλεύουν. Φαίνεται τουλάχιστον. Και δις ε, επενδύονται για την έρευνα. Όμως, τι βλέπουμε, πριν από 15 χρόνια, συγγνώμη, πριν 15 μέρες, είδαμε ότι έγιναν κάποιες έρευνες. Αλλά είδαμε ότι υπήρξαν τραγικές συνέπειες. Πού οφείλεται. το γεγονός ότι μπορεί τα οχήματα τα ηλεκτρικά αύριο να είναι ακόμα πιο επικίνδυνα από τα σημερινά οχήματα όπως έδειξαν κάποιες τραγικές συνέπειες από κάποια πράγματα. Και τελευταία ερώτηση για τον GEAR 2030 στις συζητήσεις σας. Κάντε προπτικές ε, μελέτες. Τι εννοώ. Η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κυκλοφορούν οχήματα με οδηγό και αυτόματα αυτόνομα οχήματα. Με ποιο χρονικό ορίζοντα έχετε κάνει κάποιες προβολές ε, και προοπτικές μελέτες. Ποιες είναι οι πίστες. Ε, θα έχουμε συγκεκριμένες λωρίδες για τα αυτόνομα οχήματα π.χ. Γιατί το έχω μελετήσει το θέμα. Στη ΣΥΠΑ υπάρχουν διαβαθμίσεις αν είμαστε στην κλίμακα 5, ένα αυτοκίνητο είναι αυτόνομο. Εντελώ. Εμείς στην Ευρώπη εδώ που βρισκόμαστε. Αν έχουν γίνει μελέτες από αυτόν ε, και από πλευρά επενδύσεων τι γίνεται. Επίσης, ένα ηλεκτρικό όχημα, το βλέπουμε ίσω λίγο στη ΣΥΠΑ ήδη, θα φέρει τα πάνω κάτω στις πόλεις σε ό,τι αφορά την αστιφιλία και τη συμπεριφορά ε, σε και με την ενέργεια. Το έχετε σκεφτεί. Data center χρειάζεται ένα τέτοιο όχημα, ενέργεια για να μπορεί να προχωρήσει. Αυτά τα data center που τα βάλουμε στις πόλεις θα καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Ένα αυτόνομο όχημα για να δει που υπάρχει μια λακκούβα με νερό χρειάζεται 38 εκατομμύρια, όχι, 390 εκατομμύρια δεδομένα, δεδομένα για να εντοπίσει μια λακκούβα με νερό. και δεν μέτρησα καν τα μηδενικά ε, που χρειάζονται για να εντοπιστεί ένα άλλο εμπόδιο στον δρόμο. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν να ε, λειτουργούν με ρεύμα ή με ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Τα οχήματα αυτά δεν είναι όμως τόσο βιώσιμη η κινητικότητα αυτή. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις. Θα σας δώσω όμως το λόγο για να προσθέσετε και ό,τι θέλετε εσείς σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Εσείς, από τον Κέρι 2030. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για να βάλουμε το πλαίσιο αμέσως. Τι είναι αυτή η ομάδα, είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου, όπως υπάρχουν και άλλες ε, που έχουμε και πολλά χρόνια. Και έρχεται από το γεγονός ότι ε, η Κομισιόν δεν έχει την αλήθεια διεπιφωτίσεως ε, και ζητάει βοήθεια και άλλων ανθρώπων έτσι ώστε να πάρει αποφάσεις. αυτή η ιδέα του Gear 2030, όπως και για άλλες ομάδες εργασίας, ήταν για να ε, υπάρχουν εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες ε, έτσι ώστε να καθίσουν ε, και τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να έχουν μια κοινή κατά κάποιο τρόπο συζήτηση για τις προκλήσεις, για την διακυβεύματα, για τον ορίζοντα. Δεν πρόκειται για νομοθετική διαδικασία, είναι μια διαδικασία διαλογισμού ε, την οποία χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν πάρει τις αποφάσεις της, αποφάσεις οι οποίες δια της νομίμου διαδικασίας φτάνουν και σε εσά. Η ομάδα λοιπόν ε, ολοκλήρωσε την εργασία της, το διαλογισμό της, αυτό τη σκέψη της τον Οκτώβριο του 2017. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Ντέλη, μπορώ να συμφωνήσω απολύτως μαζί σας αυξάνονται οι προκλήσεις ε, και επομένως θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, να δούμε εάν το κανονιστικό πλαίσιο είναι σωστό, αν ε, τα, οι κανόνες είναι σωστοί, αλλιώς θα πρέπει να τους προσαρμόσουμε. Η κεντρική ιδέα βεβαίως είναι ότι πολύ συχνά το ε, το ερώτημα είναι χρειαζόμαστε ένα ειδικό πλαίσιο ας πούμε για την αυτοκίνητη αυτοκίνηση στον τομέα της κινητικότητας ή θα πρέπει απλώς να ενταχθεί στην γενικότερη όσον αφορά τους, τις μπαταρίες. Έχουμε στερεά κατάσταση στην Ευρώπη, όχι, στην, όχι στο Εύρος που ε, θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική βεβαίως ε, σε σχέση με άλλους. η πρωτοβουλία αυτή, η Battery Alliance, αυτή η πρωτοβουλία θέλει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ε, ευρωπαϊκής ικανότητας ε, παραγωγής ε, των λεγόμενων σωλευτών δεύτερης γενιάς second generation batteries. Αλλά δεν είναι και αυτό ο κύριος στόχο, Ο κύριος στόχο στην ουσία είναι να υπάρχει η δυνατότητα και η γνώση για παραγωγή των μπαταριών τρίτη γενιάς. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να ε, ε, ε, αποκτήσουμε γνώση η οποία θα απορρεύσει από την εμπορευματοποίηση της δεύτερης γενεάς μπαταριών. Ναι, το, η στερεά κατάσταση υπάρχει. Δεν είναι περί αυτού ο λόγος. Απάντως δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί όσο άλλες ε, τεχνολογίες. Για τα υπόλοιπα θα αφήσω το λόγο στον συνάδελφο Έντι από την DG Connect για, τα, για τη διασύνδεση αυτοκινήτων κλπ. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία. βιομηχανία; um, Με το Gear 2030 θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί εξορισμού η ψηφιοποίηση και στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλες θα φέρει αλλαγές. Δεν μπορούμε, δεν είναι μαγική εικόνα να εξαφανιστεί. Έχουμε άλλωστε και κλιματικούς στόχους που έχουμε θέσει για τα επόμενα χρόνια, αλλά, αλλά υπάρχει αυτό το περιβάλλον το οποίο δεν θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το Kiev 2030 είναι να βρούμε εάν υπάρχουν κάποιες, ε, ε, κάποιες ε, επιφάνειες επαφής κατά κάποιο τρόπο, ε, εάν μπορούμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας σε ορισμένα σημεία. Δεν υπάρχει λόγος ε, να θεωρήσει κανείς ότι υπάρχει τοξικό περιβάλλον ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία στις ε, εκθέσεις μας. Ε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας γενικώ. Όσον αφορά τώρα τις πρωτοβουλίες για ε, μοιρασμένη χρήση αυτοκινήτου, car sharing κτλ. Κοιτάξτε, είναι πιθανό ενδεχομένως να μειωθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων, αλλά μην λησμονούμε ότι η συνολική ζήτηση αυτοκινήτων συνολικά αυξάνεται. Γιατί δεν είναι η Ευρώπη η μοναδική αγορά στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς ίσως δεν μειωθεί η παραγωγή στην αυτοκινητομηχανία έστω και αν προκύψουν κανόνες μέσω των οποίων στην Ευρώπη θα μειωθεί η ζήτηση των αυτοκινήτων. αλλά πρέπει να ληφθεί και αυτή η διάσταση υπόψη. Συμμετοχή στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου. Δεν είμαι η Δήμων περί τα θεσμικά, αλλά νομίζω ότι εμείς δεν θεωρήσαμε ότι έπρεπε να είμαστε μέρος της θεσμικής ε, ε, συζήτησης και να είμαστε ας πούμε ένα θεσμοθετημένο σώμα. Συμβολή στη συζήτηση θέλαμε να κάνουμε. The Σκάνδαλο δίζελ. Πολλής λόγος έγινε για το θέμα αυτό, όμως δεν, ε, ε, ε, και, το ζήτημα από τη στιγμή που προκύπτει η παράβιαση νόμου παράβαση νόμου δεν θα συζητηθεί εδώ, αλλά βεβαίως η Κομισιόν ήταν proactive για τα θέματα αυτά. Έχει δημιουργήσει εργαλεία ε, για τον έλεγχο, έχει τροποποιήσει ε, τα πρότυπα των ελέγχων ε, και μάλιστα τώρα θα προχωρήσει η τέταρτη δέσμη τροποποίησης για τους ελέγχους των οχημάτων. Η Κομισιόν χτες ενέκρινε και το νέο Deal for Consumers, τη νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, που θα μελετήσετε κι εσείς όταν ε, φτάσει στο Κοινοβούλιο. Παρατηρούμε τις διάφορες εκστρατείες που λαμβάνουν χώρα στις χώρες μέλη και υπάρχουν περιπτώσεις ε, ε, για τις οποίες η Κομισιόν έχει ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση. Ο καθένας όμως παραμένει ε, στα πλαίσια του, μελετά τον ανταγωνισμό, παραβιάσει σχετικά με τον ανταγωνισμό, παραβιάσει τον νόμο κλπ. Και ξεκινούν οι αντίστοιχες διαδικασίες. Όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτών των ε, εξελίξεων, ε, το είπα και στην παρουσίασή μου. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που είπα στην αρχική μου παρουσίαση. Υπάρχει και μία ε, έρευνα πάντως που έχει μελέτη συγγνώμη, που έχει ξεκινήσει από το ερευνητικό κέντρο που αφορά ακριβώς ε, το, τα όσα περιλαμβάνονται στο, στο τέταρτο πακέτο για την κινητικότητα που θα παρουσιαστεί το Μάιο. Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη μελέτη ε, για την επίπτωση της ψηφιοποίησης και της διασυνδεδεμένης οδήγησης στην κοινωνία διαδικασίες και δραστηριότητες λοιπόν που ανέφερα τώρα ή ε, και πριν ε, δείχνουν ότι φυσικά είναι μια διάσταση που μας απασχολεί πάρα πολύ αυτή της επίπτωσης της ε, ψηφιοποίησης. Yeah, on, the, on safety, um, we are actually uh, um, we are of course conscious of that. Just example. Σας δώσω ένα παράδειγμα στην τρίτη δέσμη κινητικότητας έγινε πρώτες τροποποίηση ε, του κανονισμού γενικής ασφάλειας και εκεί προβλέπονται τρεις μεγάλες ε, αλλαγές ε, οι οποίες δεν υπήρχαν στο προηγούμενο πλαίσιο. Έχουμε διάφορα όπως είναι ας πούμε η βοήθεια, η υποβοηθούμενη μάλλον αύξηση ταχύτητας και διάφορα άλλα τέτοια τα οποία αφορούν ε, την ε, οδική ασφάλεια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο εγώ, αλλά μόνο μία ερώτηση για τα data centers. Εδώ όσον αφορά αυτά τα, αυτά τα κέντρα, ε, εμείς ε, εφαρμόζουμε, θα εφαρμόσουμε και ένα μέτρο προστασίας του οικολογικού σχεδιασμού, eco-design. Ξέχασα να αναφερθώ στο θέμα των πρώτων υλών Αναφέρθηκα προηγουμένως στο γεγονός ότι λαμβάνουμε υπόψη μας όλη την αλυσίδα και ε, συμπεριλαμβανομένου και των πρώτων υλών. Εκεί συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η ανακύκλωση. Υπάρχουν πολλές ε, ε, δυνατές πηγές κοιτάμε διάφορες δυνατότητες. Ε, ε, υπάρχει στη Σουηδία και στη Σλοβακία και στην Σουηδία ε, υπάρχει κοβάλτιο το οποίο μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί. και επομένως μπορούν είτε να, ε, είτε να ξεκινήσει είτε να επανεκκινήσει η εξόρυξη κοβαλτίου. θα πρέπει να το δούμε το θέμα συνολικά των πρώτων ε, ύλων. Και ούτως ή άλλως όταν λέω ότι μας απασχολεί η διαδικασία από τις πρώτες ύλε μέχρι την ανακύκλωση, δεν σημαίνει ότι οι πρώτες ύλε οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεθούν επί ενωσιακής επικρατείας. Ναι, συνεχίζει η Κομισιόν ε, DG Move και μετά θα υποβάλω ερώτημα στην DG Connect. Ε, θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ πάνω σε τρία σημεία. Ε, το πρώτο έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στο σύστημα μεταφορών. Ε, να δούμε τι γίνεται στο αστικό περιβάλλον. Έχει γίνει ένα τεράστιο έργο μέσα σε λίγους μόνο Τον περασμένο Οκτώβριο, Νοέμβριο περίπου ξεκινήσαμε μέσα στις επιτρο... μέσα στις Επιτροπές, Επιτροπές Συστημάτων Μετακίνησης να ε, εξετάζουμε το, το τι συμβαίνει, να δούμε τι ε, εξελίξεις αναμένουμε από την ε, βιομηχανία και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των αρχών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε περιπτώσεις όπου έχουν αξία την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Όχι μόνο εμπορική αξία αλλά και δημόσιο συμφέρον. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις, να δούμε τη λειτουργικότητά τους και δεν θα σας εκπλήξει αν σας πω ότι είδαμε πως οι συλλογικές ε, μεταφορές ε, ήρθαν στην πρώτη θέση. Οι μαζικές μεταφορές, συλλογικές μαζικές μεταφορές. Αν δούμε τη λευκή βίβλο για τις μεταφορές, όσο μεγάλο και παλιό έγγραφο κι αν είναι, θα δούμε πως δεν έχουμε περιθώριο να μειώσουμε την, ε, τις μεταφορές. Ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις πόλεις είναι γεγονός ανεξάρτητα από το τι θα καίει το αυτοκίνητο. Είτε ηλεκτρικό είναι είτε καίει η βενζίνη, πάλι θα δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό μέσο αντιμετώπισης των προκλήσεων και να προετοιμάσουμε τις πόλεις έτσι ώστε να προσαρμόσουν τον αστικό σχεδιασμό στις νέες τεχνολογίες. όλη αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει με τις ε, δημόσιες αρχές ε, όμως ε, δεν έχει κάποια σύνδεση με τη βιομηχανία, δεν υπάρχει επικοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς να δούμε αυτές τις λεπτομέρειες, να δούμε τα χρονοδιαγράμματα και πώς η βιομηχανία μπορεί να μπει και αυτή στο παιχνίδι. Έπειτα σε ό,τι φορά την ε, ασφάλεια. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Όχι μόνο από νομοθετική απόψη, αλλά και στην πράξη. Να δούμε πώς ε, θα λειτουργήσει ε, όλη αυτή η εξαρτία της πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, πώς ε, μπορούμε να εξοπλίσουμε τα οχήματα, δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ρυθμίσουμε τα πάντα, όμως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα επιμέρους στοιχεία και τις επιπτώσεις που θα έχουν στους τελικούς χρήστες. Και εδώ έρχεται στο παιχνίδι και η συνδεσιμότητα. Τα συστήματα μεταφορών συμπεριλαμβάνουν και τα αυτοματοποιημένα οχήματα, τα οποία χρειάζονται επίσης ε, ασφάλεια. Και χρειάζεται λοιπόν να ανοίξει κάποια επικοινωνία ανάμεσα στα οχήματα και στα συστήματα ασφαλείας έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια. Μετά, ε, δεδομένα. Έχουν γίνει ήδη πάρα πολλά με τη σχετική οδηγία και προσπαθούμε να πιέσουμε για περισσότερη προσβασιμότητα στα δεδομένα αυτά, τα οποία δεδομένα δεν είναι απαραίτητο να φτάνουν από ε, το κοινό προς τους χρήστες, αλλά και αντίστροφα. Πρέπει να αμφίδρομη η ροή των δεδομένων έτσι ώστε να αποφεληθούν όλοι από αυτό και να οργανωθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα η ροή ανθρώπων και εμπορευμάτων. Σας ευχαριστώ. Ναι, αλλά κυρία Ντεπρέ, όσον αφορά τα δεδομένα, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Ορθώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην έκθεση καμία αναφορά στην πρόσβαση στα δεδομένα. Δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα. Εγώ υπέβαλα ένα πραγματικό ερώτημα πριν. Στην εργασία σας με τους με την αυτοκινητοβιομηχανία έγιναν προτάσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, γιατί αυτό είναι ένα πραγματικό ζήτημα και μια πραγματική ερώτηση. Το αντιμετωπίσατε, το συζητήσατε, υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία ε, προβληματισμού όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσω απαντώντας στην ερώτηση αυτή λέγοντας ότι υπάρχουν κάποιες απαιτήσει προϋποθέσεις σήμερα ήδη που εφαρμόζονται ήδη επί τη βάση της ε, οδηγίας αιτιάς δεν περιμένουμε απλώς, ε, δεν προσδοκούμε, απαιτούμε ε, ε, την πρόσβαση σε δεδομένα και την απόδοση από πλευράς βιομηχανίας κάποιων στοιχείων. Και συζητούμε λοιπόν με την αυτοκινητομηχανία έτσι ώστε, έτσι ώστε αυτός ο οποίος προμηθεύει ίδιες και παρέχει ίδιες υπηρεσίες ε, με βάση ας πούμε ε, παρόμοιες ε, περιβαλλοντικές συνθήκες και οδηγό φάντασμα, νομίζω πως έτσι το λέμε λέει η ομιλήτρια να δίνουν λοιπόν όλα τα δεδομένα όσον αφορά αυτά τα στοιχεία και, άλλα στοιχεία επιπλέον. Επομένως αυτός ο διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει. Δουλεύουμε για τη για την επιτάχυνση της διαδικασίας ε, αποδόσεως των δεδομένων και θα αφήσω μάλλον το λόγο στον εκπρόσωπο της DigiConnect. Πρόεδρος. Ναι, να μας πείτε λίγο και σε σχέση με αυτά που μας είπε και ο κύριος Μάση ποια είναι η δική σας άποψη γιατί όλα αυτά θα αποτελέσουν μια καλή βάση για τις μελλοντικές μας συζητήσεις. Ένα μόνο θα πω για το γενικό και ειδικό. Το είπε και ο Γκουέν πριν. Ο καθηγητής Μάση θα πρέπει να δώσει στην Επιτροπή Ενέργειας ε, τα, ε, του για τους ευφύς μετρητές ε, και επίσης θα μιλήσουμε για τα όσα έγιναν ε, για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια σε άλλες ε, ομάδες. Εμείς είδαμε ότι υπάρχει εγκάρσιες εξελίξεις. 5G, δεδομένα, κυβερνοασφάλεια, αλλά υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη και άλλα. Όχι μόνο η γάμα Delta Connect, είναι εσωτερική συζήτηση, αλλά και κάποιοι άλλοι από τις τηλεπικοινωνίες ε, το έθεσαν το θέμα και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα μοντέλα δεδομένων. Εμείς το συζητάμε συνεχώς το θέμα. Άρα εκεί είναι το θέμα. Generic specific. Δεν είναι και το τέλος όμως της όλης κατάστασης. Θα ακούσουμε τις νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες του Γιούνκερ ε, στα τέλη Μαΐου περίπου. Εκεί θα περιλαμβάνονται προτάσεις για την κυβερνοασφάλεια. Σκάναμε τον Σερ του Έχουμε 25 Απρίλια, έχουμε το το κινητικότητας μετά. Συνεχίζουμε και την κουβέντα μας εμείς. Το 5G. Είναι παράδειγμα, έχει ρυθμιστικές εξουσίες η Κομισιόν. Εμείς έχουμε δημοσιονομικές τόπε η ε, Κλέρ για το ΣΕΦ. Έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Και έναν διαγωνισμό έχουμε προκηρύξει. 50 εκατομμύρια για το 5G, ιδίω για την κινητικότητα. Άρα βλέπουμε λεπίδραση. Ειδικού και γενικού. Δεν θα σταματήσουμε την κουβέντα. Το κύριο 2030 ολοκλήρωσε. Όλοι συνεχίζουμε τις κουβέντες μας και τις συζητήσεις μας. Uh, uh, uh, um, και προσπαθούμε να βάλουμε και την πλατφόρμα των ε, εμπλεκόμενων φορέων, το ITS και όχι μόνο το Gear 2030 μέσα στο παιχνίδι και στις συζητήσεις αυτές. Αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε στο θεωρητικό επίπεδο, θέλουμε να πάμε και στην πράξη δεν θυμάμαι πώς το λέμε τώρα, αλλά τέλο πάντων, κάτι ψηφιακούς, διασυνοριακούς διατρόμους. Ελλάδα, επαναλαμβάνω, διασυνοριακά, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε τις δοκιμές και μετά βλέπουμε. Τι γίνεται με τα δεδομένα, πώς λειτουργεί το μοντέλο ασφάλειας, ε, συνδεσιμότητα, αυτά τα δεν βλέπουμε και τα κάνουμε δοκιμές σε πραγματικό χρόνο με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Η Ευρώπη έχει καταφέρει πολύ καλά ε, να καταφέρνει να υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, παρασχάρη μεταξύ μεταφορών και επικοινωνιών. Πολύ σοβαρή συζήτηση αυτή που γίνεται. Τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία, Gear 2003, πολλές συζητήσεις. When we start taking action and we do it in a fragmented way. Το θέμα είναι να μην υπάρχει κατακαιρματισμός. Γι' αυτό κάνω τη συλλογική προσπάθεια και με τη δική σας βοήθεια. Διάβασα την έκθεση της πρωτοβουλίας για το ITS. Αλλά είναι κατεπήγον να αναλάβουμε συλλογική δράση. Και είναι και κάτι άλλο εγκάρσιο έναντι τομεακό, κλαδικό. Και αυτό είναι ο νεοτερισμός. Έχω και κάποια ερωτήματα για εσάς. Η έκθεση σας πάντως ήταν πάρα πολύ καλή και Έχει Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουμε μία μοναδική πρόκληση. Να συνενώνουμε όλα αυτά. Ε, δύσκολο στην πράξη, αν και μπορεί να φαίνεται εύκολο στο χαρτί. Ε, ευχαριστούμε κύριε Μάσε, εσείς, για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν και θα ήθελα να τονίσω ότι κάποια από τα πράγματα που έχουν ε, γίνει, κάποιες προτάσεις είναι επικριτικές. Δεν είναι όλα υπέρ. Γι' αυτό θα είναι απαραίτητο έτσι ώστε να ε, εξασφαλίσουμε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι δηλαδή πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν ε, σκορπίζουμε τις ιδέες από εδώ και από εκεί και δεν χάνουμε την ουσία. Νομίζω πως αυτή είναι και η συνεισφορά των ομάδων αυτών, δηλαδή να κοιτάξουμε τη γενικότερη προσέγγιση, τη γενικότερη εικόνα και όσο και το αν είμαστε στο σωστό δρόμο, θεωρώ πως είμαστε σε ένα σημείο καμπής και η δουλειά που κάνουν αυτές οι ομάδες θα βοηθήσει στο να αποφασίσουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Και έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο το όχημα ε, σημαντικό. Το όχημα ε, συνδέεται και με το έξυπνο επικοινωνεί με το κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι ξεκάθαρο ε, σε ποιον τομέα ανήκει, αν, είναι στο, αν ανήκει στο τομέα της κινητικότητας, της ενέργειας, ε, είναι λίγο πολλά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ε, κοινό πρότυπο για όλους τους τομείς και να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, απομόνωση. Κάθε φορά που επιλέξαμε το δρόμο της απομόνωσης και είπαμε ότι εντάξει το, θα κάνω τη δική μου πλατφόρμα, τη δική μου προσέγγιση, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης μπαίνουν στο παιχνίδι, επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και βλέπουμε ότι αυτές οι προτάσεις, ε, οι απομονωμένες, δεν επέζησαν. Πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με όλους τους ε, σχετικούς ε, κλάδους. Πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα. Δεν ε, εταιρεία που αναπτύσσει ε, πρωτόκολλα λογισμικό και τα λοιπά να, μην μπορεί, να αναπτύξει ένα προϊόν το οποίο δεν μπορεί να συνδεθεί με τίποτα άλλο και θα είναι αυτόνομο. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε τις γενικότερες σχέσεις και η Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν άπειροι υπολογισμοί, άπειρη δουλειά που έχει γίνει που κοιτάζει ακριβώς αυτό, να μην ε, υπάρχουν προβλήματα να, ε, και σχετικά με το θέμα της ασφάλειας. Φυσικά και πρέπει να δούμε τα δεδομένα, να φροντίσουμε να μην μπορεί κάποιος να πάρει τον έλεγχο του οχήματο από απόσταση και να μην... και τα δεδομένα που λαμβάνουμε να είναι αξιόπιστα, έτσι ώστε όταν ας πούμε, το σύστημα εντοπίσει μια λακκούβα στο δρόμο να μπορεί το όχημα να την αναγνωρίσει, να την αποφύγει. Ε, τώρα, ανεξάρτητα από το αν το όχημα αυτό θα είναι ε, θα έχει οδηγό ή όχι, τον αυτόνομο, πώς θα κινείται κτλ. Μπορεί στο μέλλον, ας πούμε, η οχι Τα αυτονομο πως θα κινειται κτλ μπορει στο μελλον ας πουμε η τεχνολογια να προχωρήσει τόσο, ώστε να μην χρειάζεται εγώ να αγοράσω αυτοκίνητο, να χρησιμοποιώ μια εφαρμογή και να έρχεται το αυτοκίνητο σε μένα. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να εξετάσουμε το θέμα από ε, όλες τις ε, πτυχές. Ίσως πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως τώρα είναι σίγουρα η στιγμή να σχηματίσουμε για να χαράξουμε μάλλον την πορεία της βιομηχανίας. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η επιτυχία μας. Ε, πρέπει να επιτρέψουμε επίσης τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και νομίζω πως ε, πάνω σε αυτό έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από τις επιτροπές σας μέχρι τώρα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχιση λοιπόν της δουλειάς αυτής ε, πολύ σωστά και αυτά που είπατε για το δίκτυο 5G. Να πω και επιπροσθετώς ότι υπάρχουν πολλά οχήματα τα οποία για παράδειγμα λειτουργούν ως ε, hotspot για ασύρματο δίκτυο. Υπάρχει επικοινωνία μέσω bluetooth, μέσω ε, από όχημα σε όχημα. Υπάρχει υποδομή. Το 5G λοιπόν είναι απαραίτητο θα έχει καθοριστική σημασία και πρέπει να κοιτάζουμε λοιπόν όπως είπα και πριν όλες τις πτυχές διαφορετικά θα χάσουμε το γενικό στόχο. Ελπίζω να κατάφερα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και σας παρακαλώ αν ξέχασα κάτι ε, να μου κάνετε και άλλες ερωτήσεις να μου το επισημάνετε. Πιστεύω πως η δουλειά που κάνουν αυτές οι ομάδες είναι καθοριστική σημασίας διότι θα συγκεντρώσουν σε ε, μία πρόταση διαφορετικές πτυχές της βιομηχανίας και ακόμα και αν μια μεγάλη εταιρεία, για παράδειγμα μια από τις εταιρείες που ανήκουν στο, στις 500 ισχυρότερες. Ακόμα και αν αυτή η εταιρεία αναπτύξει μια, δικιά, μια δική της μέθοδο, πρέπει ε, για να μπορεί να την ε, εφαρμόσει, να την πουλήσει, να ε, καταστήσει δυνατή τη σύνδεσή της με όσο το δυνατόν περισσότερες άλλες τεχνολογίες. Και ε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι διαφορετικά θα χάσουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να βρεθούμε στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μασέ. Νομίζω ότι μπορούμε να σας ε, συγχαρούμε, να σας ε, χειροκροτήσουμε Connect. Ε, και Move σας προειδοποιούμε, θα παρακολουθούμε από πολύ κοντά όλα τα ε, ζητήματα αυτά και τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω εάν μπορώ να είμαι μέλος ε, σε αυτή την ομάδα εργασίας, αλλά θα σας παρακολουθούμε από πάρα πολύ στενά. Δεν το κάνω γιατί είμαι κακός άνθρωπος και γιατί θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να πάρουμε τις αποφάσεις, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μάση, είναι μετρημένος ο, ο χρόνος μας. Αυτά λοιπόν, εάν δεν έχουμε κάτι υπό τα διάφορα, σας αποχαιρετώ και στις 25 Φεβρουα... Ε, Απριλίου, συγγνώμη, στις 9 το πρωί θα τα ξαναπούμε. Α, δεν είναι Δευτέρα, δεν είναι Δευτέρα 25 Απριλίου. Ναι, Δευτέρα 9 η ώρα το πρωί, όχι, είναι Τετάρτη 9 η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ, γεια σας.